Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, έχετε κανένα πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη, συμφωνείτε να την εγκρίνουμε. Λαμπρά, να καλωσορίσω την Επίτροπο Μπούλτς για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις ε, σε σχέση με το κόρσε, δηλαδή το σύστημα αντιστάθμισης του διοξιδίου του άνθρακα και των μειώσεων εκπομπών τη διεθνού αεροπορία, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορία. Έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για απόφαση του Συμβουλίου ε, και θα δούμε τι θέση θα λάβει στον ΔΟΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά ε, τα πρότυπα και τι συνιστόμενε πρακτικέ, τα SARPS. Έχουμε δύο επιστολές που έστειλε η ΔΟΠΑ προς το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, δεν θα μακρηγορήσω όμως εγώ. Θα δώσω το λόγο στην αρμόδια επίτροπο την κυρία Βιολέτα Μπούλς για να σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απαλλαγή της αεροπορίας από τις εκπομπές άνθρακα σίγουρα είναι πρωταρχική προτεραιότητα της Επιτροπής και από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων της και φαντάζομαι ότι θα παραμείνει τέτοια ύψιστη προτεραιότητα και θα παραμείνει στο πολιτικό πρόγραμμα όχι μόνο της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των επόμενων. Μάλιστα, είμαστε προσκολλημένοι στους στόχους Συμφωνίας των Παρισίων και για να τους υλοποιήσουμε πραγματοποιούμε μια μία αναστρέψη μεταστροφή προς μια κινητικότητα με χαμηλές και εν τέλει μηδενικές εκπομπές ε, και μάλιστα μηδενικές μέχρι το 2050. Αυτός, αυτός είναι και ο στόχος μακροπρόθεσμης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου. Η στρατηγική μας ξεπερνάει τις μεταφορές και καλύπτει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οπότε το ερώτημα δεν είναι πια αν και κατά πόσο, αλλά με ποιο τρόπο. Περάμε τώρα στην αεροπορία. Είναι ισχυρός κλάδος της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ένα σημαντικό μέσο μεταφοράς. Η ανάπτυξη της αεροπορίας παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και βοηθά την περιφερειακή ανάπτυξη προσελκύοντας εμπορικέ δραστηριότητε και επενδύσει. Αλλά η ανάπτυξη για την ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αυτό ο σκοπός. Η, αεροπορία έχει και εξωτερικού παράγοντε που την επηρεάζουν που θα πρέπει να του παραβλέπουμε. Οι άμεσε εκπομπέ τη πολιτική αεροπορία είναι περίπου το 30% των συνολικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από το 2% των παγκόσμιων εκπομπών. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από την αεροπορία συμπερίληφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών από το 2012. Μέχρι στιγμής ε, το σύστημα έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα της αεροπορίας. Αυτό είναι γεγονός. Τα λειτουργικά μέτρα όπως ξεχρονισμό και η βελτίωση των ε, τεχνολογιών ε, ε, διαδικασιών και συστήματων διαχείριση ενέργεια κυκλοφορία συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών τη αεροπορία. Επίση, χάρη στι νέε τεχνολογίε αεροσκαφών, τα καθαρότερα καύσιμα και την ανανέωση των αεροσκαφών, καταφέραμε να έχουμε σήμερα 40% χαμηλότερε εκπομπέ ανά χιλιόμετρο από ό,τι το 1992. Όπως γνωρίζετε, αυτό το σύστημα, το Κορσία, σύστημα στάθμισης διοξείδου του άνθρακα και μιας εκπομπών διεθνής αεροπορίας, είναι το πρώτο ε, παγκόσμιο τέτοιο πρόγραμμα για την αεροπορία που υλοποιεί και επεκτείνει τη Συμφωνία των Παρισίων και συμβάλλει στην στρατηγική για την αεροπορία και στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. και σίγουρα χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε τις ε, εκπομπέ τη διεθνού αεροπορία. Και μάλιστα είχα την τιμή να είμαι στο Μοντρεάλ όταν ε, επετέφθη η συμφωνία. Και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και εσεί ε, προσπαθείτε εργοδός ώστε να διαφυλάξετε την περιβαλλοντική αικαιρεότητα του Κορσία. Και γι' αυτό δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και τεχνική αρρωγή για να βοηθήσουμε τις χώρες να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο, το Κορσία. Μέχρι στιγμής έχουμε τρία σχέδια αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν προσφερθεί να λάβουν μέρος εθελοντικά στην πιλωτική φάση του Κορσία μέσω της διακήρυξης της Μπρατισλάβα. Και παγκοσμίω 76 χώρες έχουν δεσμευθεί, χώρες που αντιπροσωπεύουν το 76 περίπου το 100 της δραστηριότητας της διεθνούς ε, αεροπορίας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η Ινδία, για παράδειγμα, θα εφαρμόσει το, σύστημα παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης του Κορσία, κάτι που είναι πολύ θετικό. Τούτου λεχθέντος, είναι αλήθεια ότι αυτό το σύστημα της στάθμισης των εκπομπών ειστερεί σε σχέση με τις φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάποιες απόψεις και το ίδιο ισχύει και για την αποτελεσματικότητα του Κορσία. Μόνο του το σύστημα εμπορία εκπομπών, ακόμη και με τι υψηλότερε δυνατέ φιλοδοξίε, δεν θα αρκεί για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τι εκπομπέ τη διεθνού αεροπορία. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί αν αποτύχουμε τώρα, θα ακυρώσουμε ε, πολύχρονο έργο που έχει ήδη επιτελεστεί. Βέβαια το ένα μέτρο δεν αποκλεί το άλλο, γι' αυτό σας προσκαλώ να συνεργαστούμε επ' αυτό το πνεύμα. Το Κορσία υπόκειται σε αξιολόγηση κάθε τριετία και μπορεί να αξιολογηθεί, να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί πολύ πριν το τέλος της πιλωτικής φάσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προωθεί για στιβαρούς και αποτελεσματικούς κανόνες. Η παγκόσμια συνένεση για το σύστημα Κορσία εξακολουθεί να είναι ευάλωτη όπως σας είπα, συμμετείχα στην τελική συζήτηση τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και σας διαβεβαιώ ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να έχουν ενδιασμούς ως προς ένα μέτρο που θεωρούν ως απειλή στην κυριαρχία τους και πρόσκομα στην ανάπτυξη της αεροπορικής τους βιομηχανίας, του κλάδου της αεροπορίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να συνεχίσει να διατρανώνει την πρόθεσή της να συμμετέχει στο Κορσία προκειμένου να δημιουργήσει μια δυναμική για την εφαρμογή. Οποιασδήποτε επιφυλάξεις για το Κορσία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το σύνολο της πολυμερούς διαδικασίας και τη ε, πρόοδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμή. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και ήδη εφαρμόζουμε τις, ε, τους κανόνες παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων και επαλήθευση του Κορσία ήδη από φέτος. Όπως ξέρετε, θα συνεχιστούν οι συζητήσει για επιλέξιμες αντισταθμίσει και τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα επιλέξιμα καύσιμα. Τώρα, τι επιρροή θα έχει η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση, η Ευρώπη στι συζητήσει αυτέ αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυρθεί, αποσύρει την υποστήριξή τη στο Κορσία τώρα. Ο καλύτερο τρόπο για να βελτιώσουμε το Κορσία είναι να συμμετέχουμε και να επηρεάζουμε τη διαμόρφωσή του στο Διεθνή Οργανισμό πολιτική αεροπορία. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λάβουν τα κράτη-μέλη ε, στην απάντησή του στο Κορσία και στι σχετικέ επιστολέ ευθυγραμμίζεται πλήρω με την οδηγία για το σύστημα εμπορία εκπομπών. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε διαφορέ μεταξύ του συστήματο αντιστάθμιση Κορσία και του Ευρωπαϊκού Συστήματο Εμπορία Εκπομπών. Αυτό δεν το κρύβουμε. Και γι' αυτό από τη στιγμή που θα θετηθούν από τον ΔΟΠΑ τα εργαλεία του Κορσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει μια ευρυθή αξιολόγηση του συστήματος και θα παρουσιάσει έκθεση στους δύο συνομοθέτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει με βάση αυτή την έκθεση πώς θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα αντιστάθμιση Κορσία και τι κανόνες θα πρέπει να ισχύσουν στις πτήσει εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε τρόπου να συνδυάσουμε το Κορσία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών με το τρόπο που θα συνάδει με τι ε, δεσμεύσει μα από τη Συμφωνία των Παρισίων και δεν θα υπονομεύει τι προσπάθειε του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτική Αεροπορία ε, για να βρούμε μια λύση που θα εφαρμοστεί παγκοσμίω. Αξιότιμη, Ευρω... Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε αεροπορικά με ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα. Γι' αυτό θα πρέπει η μελλοντική συμφωνία και ανάπτυξη τη αεροπορία να συνάδει με του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Και για να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από την ε, αεροπορία, θα πρέπει να αποδεθούμε σε ένα διπλό έργο. Καταρχήν, να έχουμε την πιο φιλόδοξη δυνατή συμφωνία στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορίας με την ευρύτερη δυνατή κάλυψη παγκοσμίω, χωρί όμως να υπονομεύουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών για την Αεροπορία. Και από τη στιγμή που θεωρηθούν από το ΔΟΠΑ όλα τα μέσα του Κορσία, θα ε, διενεργήσουμε μια ευρυθή αξιολόγηση του συστήματο αυτού και θα σα παρουσιάσω έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σα θέλω παρακαλώ πάντως να υποστηρίξετε την όλη διαδικασία, αυτή την θερμή έκκληση απευθύνω, να συνεργαστούμε προκειμένου και η αεροπορία μα να γίνει πιο οικολογική, με ελεγχόμενο όμως και βιώσιμο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο σχολείων ε, και ερωτήσεων. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την κυρία Γκέλιγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να κάνω μερικές ε, απλές ε, και άμεσες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Συμφωνώ μαζί σας και πράγματι αυτή η Επιτροπή συμπορεύθηκε με την ιδέα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Ενδεχομένως, ε, ε, ακόμα και μετά την αναχωρησή μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε πραγματικές φιλοδοξίες στα πλαίσια του Κορσία Κατένα, κανένα στο κοινοβούλιο δεν είπε ότι με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Παρόλα αυτά, όμως, ε, συμφωνήσαμε να συμμορφωθούμε. Ήμασταν πάντοτε απόλυτα σαφείς. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο, ε, λιγότερα σαφή. Είπατε ότι το Κορσία βασίζεται στη στρατηγική των Παρισίων. Διαφωνώ απόλυτα. Δεν νομίζω, γιατί οι δεσμεύσει που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Παρισίων δεν μπορούν να, να γίνουν σεβαστές μέσω του Κορσία. Είπαμε ότι θα πρέπει να επιφέρουμε και ορισμένες ε, βελτιώσεις. Πραγματικά νιώθω κάποια σύγχυση. Αυτή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις δράσεις που αφορούν την αλλαγή του περιβάλλοντος. Θα ήθελα ευγενικά να πω ότι μάλλον κάνουμε λάθος, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, α το δεκτούμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι. Πραγματικά όμως δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσαμε να μην υποβάλουμε επιφυλάξεις μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο θα σημάνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε τα περιβαλλοντικά μέτρα στο Κορσία και ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Με άλλα λόγια, στην ουσία δεν έχουμε το δικό μας ITS ε, ε, για την αεροπορία δεν είπατε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα σας ζητούσα λοιπόν να μου πείτε για αυτό λόγο, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ακόμα βεβαιότητες, πράγμα που αναγνωρίσατε και εσείς για το Κορσία, τουλάχιστον για τα θέματα τα περιβαλλοντικά, για ποιο λόγο δεν ενθαρρύνουμε αυτές τις επιφυλάξεις ως Ένωση έχουμε ένα διαφορετικό νομικό καθεστώ, αλλά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εκφράζουμε επιφυλάξεις. Θα ήθελα λοιπόν με σαφήνεια να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επιτρέψα μου να αναφερθώ η πρόσφατη εμπειρία μου στην Κίνα. Όταν μιλήσαμε για το Κορσία, μας κοίταξαν και είπαν ότι στην ουσία δεν θα κάνουμε τίποτα. Στο Λονδίνο μίλησα σε μία διοργάνωση όπου συμμετείχαν ε, πολλοί από το τομέα της ε, αεροπορίας ε, των εναέριων μεταφορών και ήταν ξεκάθαρο ότι είναι πρόθεση όλων να μην συνεχίσει να εκφράζει επιφυλάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν γιατί δεν θα το κάνουμε αυτό μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριος Ντάς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Βεβαίως συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν, ειδικά με το ότι οι φιλοδοξίες σε ό,τι αφορά το Κορσία δεν είναι επαρκής για να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών μετά από την διάσκεψη του Παρίσιου. Βεβαίως ε, είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι όταν πρόκειται για το κλίμα και εδώ υπάρχει μία απλή αρχή ότι η αναθεώρηση που θα κάνει η Επιτροπή δεν θα πρέπει να προδικάζεται. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης. Νιώθω κάποια σύγκυση. Προτείνατε να υπάρξουν επιφυλάξεις. Ίσως κάνω και λάθος. Τα Εγώ σύμφωνο απόλυτα ότι είναι απαραίτητο να εκφραστούν επιφυλάξεις, και θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να διευκρινίσετε την άποψή μας γι' αυτόν. Δεύτερον, γιατί περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Η 1η Δεκεμβρίου είναι πρώτον πυλώνα. Ε, το θέμα ε, είναι ότι καθυστερούν πολύ οι αποφάσεις για την επιφύλαξη και ε, θα είναι ε, σχεδόν αδύνατον να εφαρμοστούν όλα αυτά. Θα ήταν δυνατόν να κυρωθεί αυτή η απόφαση στο Συμβούλιο. Είναι εφικτό αυτό μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Ντεμεσμέκερ. Παρακαλώ. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των ερωτήσεων, θα ήθελα να η απάντηση να δίνεται μετά από την ερώτηση. Υπάρχει μια επιστολή από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι γνωρίζουμε, η Επιτροπή κινητοποιείται και πριν από την 1η Δεκεμβρίου θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να τα ακούσουμε αυτό και μετά συνεχίσουμε, γιατί στην ουσία τίδενται οι ίδιες ερωτήσεις. Ωραία. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε μια διαφορετική ερώτηση εσείς. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει μόνο μία ερώτηση. Ο κύριος Ντέμας Μάκερ, αν θέλει να πάρει το λόγο και μετά θα δώσω και πάλι το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγιναν μέχρι τώρα. Κύριε Ντέμας Μάκερ, θέλετε να διατυπώσετε την ερώτησή σας αφού πάρει το λόγο η Επίτροπος ή θέλετε να μιλήσετε τώρα. Ήθελα να ακούσω πρώτα αυτό που έχει να πει η Επίτροπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ωραία. Περιμένει λοιπόν και ο κύριος Ντεμασπάκερ να ακούσει την απάντηση που έχει να δώσει η Επίτροπος. Ας ακούσουμε λοιπόν την απάντηση και μετά θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Ωραία. Πρέπει να, μετράω, να μετρήσω τα λόγια μου. Γιατί το θέμα αυτό το συζητάμε πολύ συχνά και όπως είπα πολλές φορές υιοθετήσαμε την πρόταση η οποία σαφώς αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Κορσία και του NETS. Πιστεύω ότι οι χώρες μέλη θα αναφερθούν στις διαφορές αυτές μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Ε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η συζήτηση και θα έχουμε άμεση εμπλοκή με τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο και βεβαίως θα κοιτάξουμε τις αναλύσεις που έγιναν προκειμένου να υπάρξει εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι από το 21 μέχρι το 35 Το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα καλύψει 956 εκπομπές. Αν κοιτάξουμε το σύστημα Κορσία την ίδια περίοδο, θα αφορά 2.711. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για να υιοθετήσουμε το σύστημα Κορσία και καταλαβαίνω βεβαίως τη δική σας απογοήτευση. Θα θέλαμε να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα για να μπορέσουμε να δεσμευτούμε. Αλλά η ρήπαση δεν έχει σύνορα και για μένα είναι μεγάλο το κίνητρο να υπάρξει δέσμευση στις υποχρεώσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια παγκόσμια επίδραση. Είπατε ότι η Κίνα είπε ότι δεν θα συμμορφωθεί. Εγώ θα πρόσεχα πριν κάνω τέτοιου είδου δηλώσεις. Η Ινδία είχε σοβαρές αντιρρήσεις και τώρα βλέπουμε ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα από πλευράς της Ινδίας. Αν η Κίνα κάνει ένα βήμα, βεβαίως θα το κάνουμε τον δικό τους τρόπο και μόνοι τους, αν η Ρωσία επανεξετάσει την άποψή της, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε συγκεκριμένα παραδοτέα στην, ε, σε ό,τι αφορά το κλίμα. Ποτέ δεν είπα ότι ανεφόρον θα δεσμευτούμε. Ζητάω από το Κοινοβούλιο να συμπορευτεί μαζί μας μέχρι το 2021 για να δούμε πώς θα πορευτούμε, πόσες χώρες θα ενταχθούν σε αυτή την πάση. Ξέρετε ότι προσεγγίζουμε τις 90. Για διοικητικούς θα έλεγα, τεχνικούς λόγους, η Κίνα θέλει να αποχωρήσει από τον κατάλογο της εθελοντικής συμμετοχής. Ελπίζω ότι θα επανέλθουν. Και πραγματικά ελπίζω ότι και η Ινδία θα ενταχθεί, θα συμπορευτεί ε, πλήρως γιατί υπάρχει σε ε, μηνιαία βάση μια, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που αφορά το κλίμα. Και πάλι δεν θα δεσμευτούμε ανεφόρων, αλλά εάν υπάρχει κάποια ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία υγιή παγκόσμια συμφωνία, αυτό αυτό θα συμβάλλει πολύ περισσότερο από το ευρωπαϊκό ETS, ε το σύστημα εμπορία. Συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου από το κλίμα για να μπορέσουμε να ε, συμβάλλουμε στο να συμπορευτούν αυτοί οι δύο μηχανισμοί. Ξέρω ότι θα επικοινωνούμε μαζί σας πριν κάνουμε οποιοδήποτε ε, βήμα. Ξέρω βεβαίως τα συναισθήματα που προκαλεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, μακάρι να μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε καθαρό αέρα για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να το πούμε εάν δεν υπάρξει μια παγκόσμια συμφωνία, μια παγκόσμια δέσμευση ή ε, ρήπανση θα αφορά και τον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρο. Okay. Thank you. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Δημερσμάκερ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Κυρία Επίτροπε, ακούσαμε ότι είστε πάρα πολύ συνετοί. Ε, μιλάτε βέβαια σαν την πυθία, σαν να βρισκόμαστε στο μαντίο των Δελφών. Ε, πάντως, οι προλαλήσατες, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών ασχολήθηκαν επανειλημμένως με το θέμα αυτό. Όπως είπατε, ο τομέας πολιτικής αεροπορίας ευθύνεται για το 2% περίπου των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίω ε, και αντιπροσωπεύει το 3% των ευρωπαϊκών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε είναι σημαντική η συνεισφορά της πολιτικής αεροπορίας για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Πάντως, ε, αυτό που είναι προφανές είναι ότι ε, εννέα μέρες πριν την καταληκτική προθεσμία εξακολουθεί να χρονοτριβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο το ίδιο να κολλησιεργούν. Γιατί λοιπόν αυτή η καθυστέρηση. Αν την 1η Δεκεμβρίου δεν θα καταθέσουμε επιφυλάξεις για τα πρότυπα και τις συνιστόμενες πρακτικές του Κορσία, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών θα υπονομευθεί. Θα υποσκαφθεί από το Κορσία το σύστημα της εκπομπών. Και για μας δεν είναι παλιδρόμηση αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι το σύστημα Κορσία δεν προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Κύριε Επίτροπε, είπατε επίσης ότι δεν θα δεσμευτούμε ανεφόρων ή πάση θυσία. Αλλά παρόλα αυτά δεν σας βλέπω και πολύ αποφασιστική. Γιατί διστάζετε και δεν ασκείτε πιέσεις. Είπατε στην αρχική σας ομιλία ότι μπορούμε να συνδυάσουμε το Κορσία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορία Εκπομπών. Εγώ αμφιβάλλω γι' αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ε, βάση με επιχειρήματα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο συστήματα, το σύστημα της στάθμισης εκπομπών και το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά. Ευχαριστώ κύριος Γκερμπράντη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι ότι βρίσκομαι και εγώ στην ίδια σύγχυση με τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Για μένα το όλο σύστημα και όλη η διαδικασία του Κορσία είναι σαν να πλέουμε μεταξύ σκύλας και χάριδης. Είμαστε μεταξύ δύο κακών, γιατί η έγκριση του Κορσία είναι απόλυτα ανεπαρκή για να μα επιτρέψει να υλοποιήσουμε του στόχου τη συμφωνία των Παρισιών. Απ' την άλλη, αν δεν συμβάλλουμε στο Κορσία, αν απομακρυνθούμε, ίσω απάδουμε ακόμη περισσότερο από του περιβαλλοντικού μα στόχου. Οπότε είναι δύσκολη αυτή η συμφωνία και η επιλογή μεταξύ σκύλα και χάριδης ουσιαστικά. Τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται στο Κορσία θα πρέπει να έχουν μια ενιαία φωνή και θα πρέπει πριν την 1η Δεκεμβρίου να συντονιστούν τα κράτη-μέλη υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφαθούν με ενιαία φόνη και να εκφράσουν την διαφωνία τους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται τώρα το σύστημα Κορσία. Γιατί αν αφήσουμε το Κορσία να συνεχίσει έτσι, πολύ φοβάμαι το δικό μας σύστημα εμπορίας εκπομπών ποτέ δεν θα μπορέσει να συμπορευθεί με το Κορσία. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές μου τις απορίες. Δεύτερο σχόλιο. Αφορά περισσότερο τις αερομεταφορές. Αλλά στο σημείο αυτό και οι πολιτικοί μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο. Κάτι που πραγματικά αδυνατό να καταλάβω είναι γιατί ο τομέας αποποιείται των ευθυνών του. Γιατί ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και λέει ότι το μόνο μοντέλο είναι η ανάπτυξη, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε α, μαγειρικό λάδι, αλλά δεν αρκεί για να έχουμε καθαρά καύσιμα για την αεροπορία. Οπότε ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας η πολιτική αεροπορία γιατί ξέρει ότι ποτέ δεν θα παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Αυτό όμω είναι ένα στίχημα που κάνουν η αρμόδια των μεταφορών που δείχνει όμω κάποια ανευθυνότητα. Γιατί δεν ανεπομίζεται τι ευθύνε του και ο κλάδο πολιτική αεροπορία. Έχουμε 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο επιβάτε στι αερομεταφορέ και μάλιστα την επόμενη 15 ετία θα διπλασιαστεί αυτό ο αριθμό. Θα φτάσουμε στα 8 δισεκατομμύρια επιβάτε. Γιατί ο κλάδο λοιπόν δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία ζητώντα ένα ευρώ από κάθε επιβάτη, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το χρόνο θα μαζεύει και μέσα σε μία 15 8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα μαζεύει για να δημιουργήσει ένα σύστημα σύστημα καινοτομία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί ε, ο τομέα αεροπορία, αναπτύσσοντα, σχεδιάζοντα και κατασκευάζοντα καθαρά αεροσκάφη. Μόνο με ρηξικέλευτε τεχνολογίε θα το επιτύχει. Μόνο με την επένδυση τεράστιων κονδυλίων στην καινοτομία θα το καταφέρει. Και αυτό δεν μπορεί να προέλθει από το δημόσιο τομέα μόνο. Θα πρέπει να προέλθουν τα κονδύλια αυτά και από τον ιδιωτικό κλάδο. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν αναγκάζουμε εμεί τον τομέα με περισσότερες πιέσεις για να βαδίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να μην θέσουμε τον κλάδο πρώτων ευθυνών του ε, και να τους ε, επισημάνουμε ότι τελική ανάλυση δεν θα είμαστε τόσο αδύναμοι όσο πιστεύουν πως είμαστε. Ευχαριστώ κύριο Σέικχοουτ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. μπορεί να είναι λίγο βαρετό, αλλά φαίνεται ότι όλοι τα μέλη τη Επιτροπή Περιβάλλοντο έχουν τον ίδιο προβληματισμό και τι ίδιε απορίε. Εγώ νόμιζα ότι τα πράγματα κάπω ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ανάλυση των προτύπων και συνιστόμενων πρακτικών που έχουν ολοκληρωθεί γιατί άλλα εκκρεμούν, εξετάζοντας όμως τα SARS που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς την περιβαλλοντική αικαιρεότητα του Κορσία. Γιατί δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη οι κανόνες αντιστάθμισης. Επίσης δεν ορίζονται τα εναλλακτικά καύσιμα επαρκώς. Και είναι σημαντικοί οι κανόνες και για την αντιστάθμιση, για τη στάση που θα ακολουθήσουμε στο Κορσία. Οπότε οι διατάξει δεν είναι ακριβώς ακόμη σαφεί και δεν γνωρίζουμε πότε το Κορσία και αν θα έχει την απαραίτητη περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Κάτι που είναι απαραίτητο για να κρίνουμε κατά πόσο θα εφαρμόσουμε το σύστημα εμπορία εκπομπών για όλε τι πτήσει ή όχι. Δεν έχουμε ακόμη τα στοιχεία για να το κρίνουμε. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να υποβάλλετε επιφυλάξει. Αυτέ οι επιφυλάξει ε, ε τουλάχιστον μια πρόταση ήδη βρίσκεται επιτάπητος. Αλλά υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας. Τυπικά, ακόμη, αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου δεν έχει τεθεί τυπικά, δεν έχει υποβληθεί, δεν έχει παρουσιαστεί ε, επίσημα στο Συμβούλιο, αν και όλοι τη γνωρίζουμε, εμέσως όμως είναι κοινό μυστικό, αλλά η πρόταση αυτή, αλλά επίσημα δεν μας την έχει ακόμη υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που είναι γελίο, γιατί ε, βλάπτει τη διαφάνεια και θα πρέπει να αλλάξει πάρα αυτά αυτή η κατάσταση. Επίσης, τα ΣΑΡΠΣ, τα πρότυπα και συνιστόμενες πρακτικές συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο. Γιατί χρειάστηκε τόσο καιρό για να καταλήξουμε σε μια πρόταση για την απόφαση του Συμβουλίου. Και έχουμε μόνο την 1η Δεκεμβρίου, οπότε θα πρέπει να ανασκουμποθούμε, να καταλήξουμε σε εκείνη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το χειρότερο θα είναι ο καθένα θα τραβήξει την πορεία του και μερικέ χώρε να υποβάλουν επιφυλάξει και άλλε όχι. Αν θέλετε να μα χρηστεύσετε, αυτό να κάνετε, αυτή τη στρατηγική να ακολουθήσετε. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλατε κάτι τέτοιο. Τώρα όμω από τι απαντήσει σα έχω την αίσθηση ότι ναι, υπάρχει όντω κάποιο κείμενο που προτείνει μια θέση του Συμβουλίου, αλλά ουσιαστικά μετά από αυτό δεν έχετε καμία άλλη φιλοδοξία. Έχετε βγάλει το κείμενο και ελπίζετε ότι 28 χώρες που ξέρουμε πόσο δύσκολα φτάνουν σε κοινή θέση, σε αυτή την περίπτωση θα συμφωνήσουν ως διαμαγείας χωρίς αφής καθοδηγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ περίμενα μια στρατηγική από εσά για το πώς τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν στην κοινή θέση του Συμβουλίου ότι έχετε σοβαρέ επιφυλάξει για την περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Θέλετε ισχυρή φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αυτό περίμενα από εσά και τώρα λέτε ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πρέπει να μετρήσω τα λόγια μου, δεν ξέρω ακριβώ τι να κάνω. Ε, οπότε η έκβαση θα είναι μια διχασμένη Ευρώπη. Και ό,τι και αν γίνει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το Κορσία θα φανούμε αδύναμη. Και αυτό με εκπλήσει. Γιατί αυτή η αλλαγή στρατηγική. Ε, εξακολουθούμε να επιδιώκουμε ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι θα κάνουμε ώστε να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή θέση πριν την 1η Δεκεμβρίου. Και ελπίζω να προτάξουμε αυτή την επιφύλαξη που όλοι διαπιστώσαμε. Αυτά προ το παρόν. Στη συνέχεια των συζητήσεων θα υποβάλω και άλλε ερωτήσει, αλλά προ το παρόν αυτά είναι τα κεντρικά ερωτήματα. Αυτή ήταν η ευκαιρία σα, Δεν θα έχετε δεύτερη για υποβολή ερωτήσεων. Καλώ σα ευχαριστώ. Και τώρα η Επιτρόπο για να απαντήσει. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, ε, εγώ είναι που μπερδεύομαι και τελώ σε σύγχυση, γιατί όταν ε, ακούω τα σχόλιά σα είναι σαν να ε, μην νιώσετε ότι συμμετείχατε από την αρχή στη διαδικασία. Και αυτό με μπερδεύει, γιατί όντω θα πρέπει να διαλέξω προσεκτικά τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε ότι από την αρχή συνεργαστήκαμε από την πρώτη μέρα και είχαμε πει με σαφήνεια ότι δεν είμαστε υπέρ των επιφυλάξεων, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές που θα τις επισημάνουμε. Ποιες είναι οι διαφορές του ETS και του Κορσία. Εμένα με μπέρδεψα τα σχόλιά μου. Εσείς με μπερδέψατε με τις δηλώσεις σας. Γιατί φαίνεται ότι ζούμε σε παράλληλους ε, ε, αλλά παρόλα αυτά από την πρώτη στιγμή μου σαφέστατη στην επικοινωνία μας και είπε ότι θέλουμε μια παγκόσμια συμφωνία, γιατί μια παγκόσμια συμφωνία θα έχει πολύ περισσότερα ωφέλη από μια περιφερειακή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα δεν θα υποβάλουμε επιφυλάξεις, γιατί υποβάλλουμε τι τις διαφορές, παρουσιάζουμε τις διαφορές. Έχετε λάβει τα έγγραφα, βλέπετε τι προτείνουμε. Ποια είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια είναι η πρόταση του Συμβουλίου τα έχω χαμένα πια μετά από τα σχόλια που άκουσα. Ίσως αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Έχουμε τα ίδια έγγραφα μπροστά μας. Στηριζόμαστε στα ίδια έγγραφα. Γιατί έτσι θα διαφυλάξει την ομοθεσία μας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών μας. Και αυτό λέει και η πρόταση του Συμβουλίου. Και σε αυτό θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει. Εγώ ζήτησα την υποστήριξή σας και τη συμπαράστασή σας και ζήτησα να πιέσετε κι εσείς όπου μπορείτε, ώστε όλο και περισσότερες χώρες να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση μέχρι το 2021. Αν δεν συμφωνείτε με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, είπαμε θα επανέλθουμε και θα αποφασίσουμε για το τι, ποιο σύστημα θα διαλέξουμε, το ETS ή το Corsia. Αλλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει ότι στα μέσα δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Το πιο σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων είναι μπροστά μα. Θα γίνει του χρόνου το Μάρτιο το πιο κρίσιμο τμήμα των διαπραγματεύσεων. Δύο από τα τρία σημεία έχουν συμφωνηθεί την περασμένη εβδομάδα και ένα ακόμη αναμένεται και εκρεμεί μέχρι την Άνοιξη. Και πάλι θα είμαι σαφής. Είμαι κατά της υποβολής επιφυλάξεων. Είμαι υπέρ της παράθεσης των διαφορών και στο Συμβούλιο και στο, στο, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για να καταλάβουν και τα μέλη του ΔΟΠΑ υπό ποιου όρους μπαίνουμε στη συμφωνία. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δείξει αδυναμίες, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρωτοστατήσει στη διαδικασία αυτή, τότε πολύ πιθανόν να μην ευοδοθεί όλη η προσπάθεια. μπορούμε για πολλούς και διάφορους λόγους να υπαναχωρήσουμε, όπως έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείες προς το παρόν. Να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρα. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, υπέρ της πυθού και υπέρ του να δείξουμε ε, πώς με την ανάπτυξη της αεροπορίας, γιατί θα υπάρξουν χώρες που θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροπορίας, ε, γιατί τώρα αρχίζουν να διαμορφώνουν ε, μεσαία τάξη και η μεσαία τάξη θέλει ε, να αρχίσει να ταξιδεύει και γνωρίζετε για ποιες χώρες μιλάω, για την Κίνα, για την Ινδία. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ιδιαίτερα για τις νέες τεχνολογίες και θέλουμε να συγχρηματοδοτήσουμε το σχέδιο για τα υβριδικά αεροπλάνα, για να έχουμε σε τελική ανάλυση αεροπλάνα που δεν θα ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Ηλεκτροδότηση και άλλα συστήματα υβριδικά για την, προώθηση, έτσι θα προχωρήσουμε. Θέλουμε να μειώσουμε στην Ευρώπη τον αντίκτυπο της αεροπορίας στηρίζοντας τρένα υψηλής ταχύτητας σε αποστάσεις μέχρι 500-600 χιλιόμετρα. Και θέλουμε να μειώσουμε την ανάγκη ε, των αερομεταφορών. Σε ό,τι φορά όμως το σύστημα, το πρόγραμμα για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, θέλω να νιώσω τη συμπαράστασή σας για να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις με πυγμή, αλλά και την έντιμη δέσμευση για μια παγκόσμια συμφωνία. Και πάλι τα στατιστικά στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Από μόνοι μας ε, και προωθώντας μόνο το σύστημα εμπορίας εκπομπών, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ ε, πιο ασθενή από μια παγκόσμια συμφωνία. Ακόμη και αν δεν είναι η παγκόσμια συμφωνία 100% συμβατή να ικανοποιεί τι προτάσει μα. Πάντω έτσι θα έχουμε την αξιοπιστία για να συνεχίσουμε να προωθούμε την, τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα. Εγώ είμαι υπέρ της απαλλαγής των, με, ε, μεταφορών από τον άνθρακα, από τις εκπομπές άνθρακα. Έχουμε κάνει πολλά και θα συνεχίσουμε. Είδατε στο, στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ότι ε, μεγάλη πρόοδο συντελέστη. Ε, και τώρα η ναυτιλία είναι πιο φιλόδοξη από την αεροπορία. Και θέλουμε και ο Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Ελευθερία να μιμηθεί το παράδειγμα του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Πάντω ελπίζω να έχετε τι σωστέ πληροφορίε, τα σωστά έγγραφα και με βάση τα ίδια έγγραφα να συζητούμε, γιατί από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε η όλη σύγχυση. Και γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να μετράω τα λόγια μου και να, λέω, να είμαι προσεκτική σε αυτό που θα πω, γιατί μερικέ φορέ δεν καταλαβαίνω καθόλου τα σχόλιά σα. Και ζητώ συγγνώμη. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρελε. Περάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, προσοχή που δίνεται από πλευρά τη Επιτροπή στο θέμα των εκπομπών που προέρχονται από τι εναέριε μεταφορέ. Όταν μιλάμε για κλιματικέ αλλαγέ, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, οι βασικοί φορεί, οι βασικοί εμπλεκόμενοι μιλάνε για το ότι πλησιάζει ο καιρό, πιέζει ο χρόνο για, την, ε, ε, για να περάσουμε στη φάση που θα υπάρχουν πλέον εκπομπέ άνθρακα. Στην τριμερή συνάντηση επιτροπή στη Λουμπλιάνα άκουσα χθε αυτά που είχαν να πούν ε, οι εμπειρογνώμονε για την επανάσταση των μεταφορών που προετοιμάσει στον τομέα μεταξύ των άλλων των εναέριων μεταφορών. Θα πρέπει να κινηθούμε σε πολλά μέτωπα και ενδεχομένω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ηλεκτροϊκά αεροπλάνα, υβριδικά αεροπλάνα και θα μειωθεί η προσπάθεια για αποφυγή μόνο άνθρακα. Θα χρειαστούν όμως περισσότερα χρόνια. Οι, οι, οι μηχανισμοί σε ό,τι αφορά το Κορσία με απασχολούν. Δηλαδή με απασχολεί το θέμα του εθελοντικού χαρακτήρα στον οποίο αναφερθήκαμε. Θα χρειαστούν 21-25 χρόνια κατά την άποψή μου προκειμένου να υπάρξει αυτός ο εθελοντικός χαρακτήρας. Κατά την άποψή σας θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τους ε, ρυθμούς. Ε, δεν ξέρω αν αυτό διευκολύνει τη θέση σας, αλλά σε κάθε περίπτωση ήθελα να σας κάνω αυτήν την ερώτηση. Ο κύριος Σολίνο. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ένα τμήμα της σύγχυσης που δημιουργήθηκε έχει σχέση με το τελείως διαφορετικό ύφο της πρώτης σας ομιλίας και των απαντήσεων που ακολούθησαν στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Γιατί στην πρώτη σας παρέμβαση, που πολύ φοβάμαι ότι δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Ε, εκφράστε την ανησυχία σας με τον ασταθή χαρακτήρα, τον εθελοντικό χαρακτήρα του Κορσία, τον πρωτόλιο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ανταπόκρισης και μετά, απαντώντας τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, στη δεύτερη σας ε, παρέμβαση, ήσταν πιο αποφασιστικοί. Είπατε θέλουμε συντονισμένη απόφαση, θα πρέπει να έχουμε νέα φωνή για να είμαστε καλοί διαπραγματευτές παγκοσμίω και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό όμως ε, θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στα έργα και να στηρίζεται από επιχειρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχαν μεγάλες φιλοδοξίες για όλα τα μέσα μεταφοράς, για τις οδικές και τις οδοδρομικές μεταφορές και δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, εκτός την αυτιλία ή την αεροπορία. Γι' αυτό όμω και για να επιτύχουμε του φιλόδοξου στόχου μα θα πρέπει να έχουμε μια σαφή στρατηγική γραμμή και μια εναλλακτική λύση. Τι μπορούμε εμεί, ω ευρωβουλευτέ, ε, και μάλιστα ε, μετά τη συζήτηση αυτή πολύ θα με ρωτάνε στην πατρίδα μου. Εγώ πώ μπορώ ω ευρωβουλευτή να εγγυηθώ τη συμφωνία των κρατών μελών ώστε να έχουμε μια ισχυρή στεναρή φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να έχουμε μια ενιαία θέση και παγκοσμίω. Και Μιλήστε για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τελικά οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι συμμαχός μας στη διαδικασία αυτή, ναι ή Sorry. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αξιολόγηση του Κόρσια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να το διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή, καθώ και το κείμενο του Κοινοβουλίου. Εμεί θεωρούμε ότι η Κόρσια είναι πάρα πολύ αδύναμη ακόμα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 100% σε αυτά που θέλουμε και που επιθυμούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η τόνη διοξιδίου του άνθρακα στους οποίους αναφερθήκατε ε, είναι κάτι ασαφές, διότι ασαφείς είναι και οι κανόνες. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η σαφήνεια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πιο προσεκτικοί στις λέξεις που επιλέγετε για την προσθέμενη αξία του Κόρσια. Είμαστε ακόμα στην αρχή, όμως δεν έχουμε προχωρήσει μακριά από αυτήν την αρχή και γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ως ε, Ευρωπαίος νομοθέτης ε, να περιοριστούν τα δικαιώματά μας. Και πράγματι είμαστε κάπως μπερδεμένοι διότι δεν έχουμε το κείμενο. Γιατί όμως δεν έχουμε το κείμενο. Εσείς ε, μας ρωτήσατε γιατί δεν το διαβάσαμε και εμείς σας απαντούμε ότι δεν το λάβαμε ποτέ, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να το διαβάσουμε. Και θα ήθελα λοιπόν να μην πέφτουμε σε, τέτοιες, ε, σε τέτοιο επίπεδο. Ε, δεν γίνεται να μην λαμβάνουμε τα κείμενα εμπρόθεσμα. Έχουμε την απέτηση να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει. Αλλά για να γίνει αυτό, ε, σίγουρα γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και αυτό ε, λόγο. Είμαστε συνομοθέτες. Το νομικό μέσο το οποίο έχετε επιλέξει με αυτές τις ε, διαφορές... Αν το θεωρείτε σωστό, τότε μπορούμε να το προχωρήσουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να κολλησιαργούμε. Χρειάζεται να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι ε, σωστό, το νομικό μέσο να είναι επίσης κατάλληλο και τότε θα ε, προχωρήσουμε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, η συζήτηση που θα γίνει με τα κράτη-μέλη θα έχει και αυτή αποτελέσματα. Θα γίνουν ε, σχόλια και προτάσεις για το ποιες βελτιώσεις επιδέχεται το Κόρσια. Ε, στο Παρίσι επίσης έχει υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία από όλους μας και αυτό λοιπόν σας παρακαλώ είναι επίγον να συνομιλήσετε με τα κράτη-μέλη χωρίς περιστροφές. αν δεν επιλεγεί ένα νομικό μέσο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, το οποίο θα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να αποφασίζει αυτόνομα, τότε θα ε, επισέλθουμε σε θεσμική κρίση. Καμία κομισιόν, κανένα κράτος μέλος και καμία διεθνής συμφωνία δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρώσει την ε, συμφωνία χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι κάτι που το λέω χωρίς περιστροφές, εδώ ε, πρέπει να μιλήσουμε στα άτα για το τι λείπει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κούτελαν τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την επισκεψή σας και για την παρουσίαση που κάνατε. Θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα σχετικά με τον κοινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 σε ό,τι αφορά το σύστημα Κορσία και το πώς θα επηρεαστεί. Γιατί πιστεύω ότι στο ψήφισμα υπήρξε μία δήλωση ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις πλειοδοξίες μας σε ό,τι αφορά τους στόχους του 2030. Τώρα προβληματίζομαι, μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιτύχει το στόχο του 2030 χωρίς να βασίζεται σε διεθνείς πιστώσεις, πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του Κορσία υπονομεύει ε, πιστώσεις που δεν θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά τους στόχους για το κλίμα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του, της ΔΟΠΑ είναι πιο δυναμός από την, ε, αυτό της Ευρωπαϊκή Ένωση πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αποφύγει έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή του συστήματος Κορσία δεν θα υπονομεύσει το δικό μας στόχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σκεφτόμουν να μην διατυπώσω ερωτήσεις προς την Επίτροπο, σε κάθε περίπτωση άλλαξα γνώμη. Μίλαμε για κλιματικές αλλαγές. Η Ολλανδία πηγαίνει πέρα από αυτό που είπε η Ευρώπη. Όλοι οι τομείς από την γεωργία μέχρι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Τι ζητάτε όμως από την εναέρια κυκλοφορία. Ε, θα έχει δικαιώματα ε, που δεν έχουν άλλοι τομείς. Δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Εδώ στο Κοινοβούλιο θέλουμε να ζητήσουμε τα ίδια πράγματα από όλους τους τομείς. Περί αυτού πρόκειται. Τα προαπαιτούμενα που θέτουμε για άλλους τομείς είναι προαπαιτούμενα πάρα πολύ πιεστικά καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για, τις, για αυτά που επιβάλλουμε σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να καταφέρουμε να δείξουμε ότι είμαστε συνεπείς και σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να τους ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, Πρόεδρε, Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια που δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Ε, μας ε, είπατε πως ε, δεν έχουμε δείξει τόση φιλοδοξία και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επισπεύσουμε τη διαδικασία του ε, ΔΟΠΑ. Επέμονη ερώτηση. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν εθελοντικό ε, χαρακτήρα ε, στις ε, και διμερείς συμφωνίες. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούμε ήδη με κάποιες άλλες χώρες και ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες χώρες σε αυτό το κίνημα. Μετά μας είπατε για την καινοτομία. Αναφερθήκατε στα υβριδικά αεροσκάφη. Αυτό, από όσο γνωρίζω, ε, δεν είναι ακόμα προγραμματισμένο. Η ηλεκτρική ηλεκτροκίνηση προορίζεται μόνο για την τροχοδρόμηση και την προσγείωση. Ε, πόσο μακριά απέχουμε από το να γίνουν τα ηλεκτρικά αεροσκάφη πραγματικότητα. Επίσης, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιοκαύσιμα, άλγες. Τώρα, Ήδη συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το ζήτημα των εκπομπών και της καινοτομία, αλλά εσείς έχετε κάποιες, περισσο... παραπάνω πληροφορίες για το ποιες καινοτομίε είναι αυτές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και ε, σίγουρα υπάρχουν πολλά που επιδέχονται βελτίωση, όμως αυτή τη στιγμή αυτά έχουμε και πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελείωσε ο δεύτερος κύκλος ερωτήσεων. Εάν λοιπόν θέλετε κάτι άλλο, μπορούμε να το συνεχίσουμε μέρο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Πολλές ερωτήσεις ε, αναφέρθηκαν στην τεχνολογία. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι έχουμε πολλές ε, πρωτοβουλίες που ήδη τρέχουν. Θέλουμε καταρχήν να βελτιστοποιήσουμε και τη χρήση του εναέριου χώρου και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη διαχείρισή του. Και γι' αυτό ε, Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και με το καθαρή εθέρες και με νέα εργαλεία και νέους μηχανισμούς. Η Rolls-Royce ε, και οι εταίροι της ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναπτύξουν ένα σύστημα με υψηλή αναλογία υβριδισμού ε, και να ε, μπορούν να χρησιμοποιούν τα υβριδικά αεροπλάνα που θα έχουν σύστημα τέτοιο υβριδική όθησης και ελπίζω μέχρι το 2030 να ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία. Αν συμβεί θα έχουμε μια νέα γενιά αεροσκαφών. και σε επίπεδο υπηρεσιών. Και μάλιστα με μικρά σκάφη και με μη επαδρομένα ε, τέτοια υπτάμενα, υπτάμενες συσκευέ μπορούμε ήδη να έχουμε ε, μηδενικές εκπομπές είτε με υπτάμενα οχήματα είτε με drones χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αν μπορούμε να επιταχύνουμε την πρόοδο, ναι, αρκεί να έχουμε περισσότερους πόρους. Και ευελπιστούμε ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, το επόμενο ΠΔΠ, θα γίνει δεκτή το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσουμε αμέσως τα νέα μας προγράμματα. Στις μεταφορές, η απαλλαγή από τι εκπομπέ άνθρακα για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικέ είναι περίπου το 60% του συνόλου των επενδύσεών μας. Και κάτι αντίστοιχο προβλέπεται και για την αεροπορία. Ελπίζουμε λοιπόν να αναπτύξουμε και νέα τέχνητα καύσιμα, να προωθήσουμε τη χρήση βιοκαυσίμων στην αεροπορία. Βέβαια, δεν αρκούν αυτά για να καταλήξουμε σε μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2050. Χρειαζόμαστε κάτι καινοτόμο ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μα για μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2050. Θέλουμε καινοτομίε στι μεταφορέ. Γι' αυτό και προτείναμε αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία στι μεταφορέ, στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν με την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι θα έχουμε επιτάχυση και της καινοτομίας και της πρόοδου. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τα άλλα εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αεροπορία, για παράδειγμα αύξηση των φόρων ε, ή σε σχέση με άλλες, άλλα μέσα μεταφοράς. Στις 3 Σεπτεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο θα δώσει σε τρεις χώρες την προκαταρκτική έκθεση και μία διεξοδική ανάλυση όλων των φόρων σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι θα διαμορφώσουμε μια σαφέστερη εικόνα για τη θέση της αεροπορίας σε, στο γενικό πολυτροπικό περιβάλλον. Και θα έχουμε ανάλυση ανά μέσο μεταφοράς και ανά κράτος μέλος που θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο. Και Όπω θα δώσουμε στο Συμβούλιο, θα δώσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προκαταρκτική έκθεση που ήδη δείχνει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η τελική φάση αυτό του εγγράφου. Πιστεύω ότι με την προκαταρκτική αυτή έκθεση θα έχουμε μία ακόμη ευκαιρία να δούμε την κατάσταση της αεροπορίας σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγγραφο. Μπορεί εγώ να μην ήμουν καλά κατατοπισμένη. Πάντως μου είπαν ότι το έγγραφο σας είχε σταλεί στις 21 Οκτωβρίου. Ότι όλοι έχετε λάβει τη νέα εκδοχή του εγγράφου. Αυτή που ανέφερα και εγώ δηλαδή. Τονίζω και πάλι, όπως λέει το έγγραφο, ότι προτείναμε να διαφυλάξουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και να το θωρακίσουμε απέναντι σε πιθανές νομικές προσφυγές, δικαστικές προσφυγές. Αυτό το είχαμε υπόψη όταν προτείναμε αντί για επιφυλάξεις να επικεντρωθούμε στις διαφορές και να επισημάνουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ του Κορσία και του ETS και να προσπαθήσουμε να τις εξομαλύνουμε γιατί θέλουμε να συγκλίνουν τα δύο συστήματα, το Κορσία με το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Επίσης, ό,τι και αν συμφωνήσουμε τελικά, δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν το 2021, οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο για να διενεργήσουμε μια διεξοδική μελέτη αντικτύπου ολόκληρου του συστήματος, που προς το παρόν δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει σε τελική ανάλυση. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ελπίζω το Μάρτιο να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Και από τη στιγμή που θα εγκριθεί θα κάνουμε την ανάλυση και τη μελέτη αντικτύπου και φυσικά θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματά της και εσάς και το Συμβούλιο. Για να δούμε πώς προβλέπουμε την ανάπτυξη των πραγματικών των καθαρών αποτελεσμάτων του Κορσία. Αυτό θα γίνει όπως ζητήσατε και εσείς, αυτή η υποβολή της έκθεσης, της ανάλυσης. Με ρωτήσετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε έξι, έξι από τις 36 έντρες στον ΔΟΠΑ. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε να ασκήσετε πίεση στις που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στη συμφωνία. Βοηθήστε και εμά να τις πιέσουμε και να τις προσετεριστούμε. Γιατί αν καταφέρουμε και φέρουμε και την Ινδία στο πλευρό μας, πάντως ο τρόπος που επικοινωνεί η Ινδία και η δέσμευση που έχει αναλάβει για το πράσινο, για το οικολογικό θεματολόγιο μας δημιουργεί πολλές ελπίδες για την θέση της χώρας αυτής. Και μακάρι και η Κίνα τελικά να προσχωρήσει. Αν τα καταφέρουμε πιστεύω ότι θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να, πιέ, να πείθουμε τους, εταίρους μας, να εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις, να προσετεριστούμε περισσότερες χώρες. Και επαναλαμβάνω, δεν θα τηρήσουμε καμία συμφωνία. Το είπαμε ξεκάθαρα. Το είπαμε και στο Μόντρεαλ στη συνεδρίαση του ΔΟΠΑ. Το είπαμε ρητά και κατηγορηματικά. Θέλουμε μια φιλόδοξη συμφωνία για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Αλλά ας δώσουμε μια ευκαιρία σε μια παγκόσμια συμφωνία. Αυτό σας ζήτησα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, στη συζήτηση. Φάνηκε το ζωηρό ενδιαφέρον των μελών της Επιτροπής για το έργο σας και ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που σας έστειλε η Επιτροπή μας για το τι θέλουμε. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι θα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία και κάθε φορά που έχουμε κάποια, κάποιο αποτέλεσμα, κάποια εξέλιξη θα σας ενημερώνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει ήδη ο καθηγητή Ράζη. Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Οι ανακοινώσει και η ενημέρωση από του τριμερεί διαλόγου θα ακολουθήσουν την παρουσίαση του καθηγητού Ράζη. Μια και έχει έρθει ο καλεσμένο μα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, καλώ. Έχουμε την αιτήσια ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του τακτικού διαλόγου που έχουμε με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, τον καθηγητή Γκουίντο Ράζι. Καλώ ήρθατε, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασιών του ΕΟΦ ε, για το 2018 και φυσικά όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζει ο ΕΟΦ θα πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο των πολιτικών προκλήσεων και του πολιτικού τοπίου που διαμορφώθηκε μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit θα έχει σημαντικές συνέπειες και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στην ανταλλαγή απόψεων σήμερα θα καλέσω πρώτα τον καθηγητή Γκουίντο Ράζη να μας παρουσιάσει τα πεπραγμένα του ΕΟΦ και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Καλώ ήρθατε κύριε καθηγητά και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Mr. Chairman, ladies, and gentlemen, and the honor to be here before you today. Uh, I think this is the last time that I will be addressing this committee in this composition before the election next year.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 Μα βοηθήσει να προχωρήσουμε χάρη της προστασία της δημόσιας υγεία και της υγείας των ζώων. Και φυσικά το πρώτο θέμα της ομιλίας θα είναι οι προετοιμασίε μας για το Brexit. Φυσικά μας ενδιαφέρει η συνέπεια του Brexit στη δημόσια υγεία. Έχουμε αναλύσει το πιθανό αντίκτυπο του Brexit στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και εργαζόμαστε συχνά και έχουμε στενή στενό συντονισμό με τους κατόχους αδειών εμπορίας φαρμάκων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ε, υπόνοιες ότι μπορεί να επηρεαστεί η προμήθεια. Και μάλιστα το σχέδιο συμφωνία αποχώρησης που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα προβλέπει μεταβατική περίοδο 21 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας το κοινοτικό κεκτημένο για τα φάρμακα θα συνεχίσει να ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, μέχρι να υπογραφεί, εμεί θα συνεχίσουμε τον πραγματισμό μα υπό την υπόθεση ότι οι κάτοχοι αδειών εμπορίας θα πρέπει να είναι έτοιμοι μέχρι τις 30 Μαρτίου του 2019. Και με αυτό το σενάριο, για 31 ακόμη φαρμακευτικά προϊόντα, 19 για ανθρώπινη κατανάλωση και 12 κτηνιατρικά, έχουμε προβληματισμό και φοβούμαστε ότι θα υπάρχουν κάποια προβλήματα με την προμηθεία τους μετά το Brexit. Και φυσικά προσπαθούμε με τους κατόχους με τους, με τους φορείς παροχής αδειών να, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και στις επιστημονικές μας επιτροπές θα εξετάσουμε διάφορα μέτρα μετριασμού καθώς και τις συστάσεις για πιθανές θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις, για εναλλακτικές θεραπείες δηλαδή που ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ασθενείς σε περίπτωση που τα φάρμακά τους δεν θα είναι διαθέσιμα. Το δίκτυό μας μάλιστα ετοιμάζεται για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και όλα τα φάρμακα για τα οποία ήταν εισηγητής ή συνεισηγητή του Ηνωμένου Βασίλειου σε μια συγκεντρωτική διαδικασία έχουν μεταφερθεί σε νέους εισηγητές και συνεισηγητές από τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των δύο χωρών Ισλανδίας και Νορβηγίας. Και τα κράτη-μέλη έχουν αναβαθμίσει και την ικανότητά τους και τις δυνατότητές τους. Τώρα, για τον ΕΟΦ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες. Ε, το σίγουρο είναι ότι σε πέντε μήνε από τώρα θα βρισκόμαστε στο Άμστερνταμ και η προετοιμασία τόσο του ενδιάμεσου κτηρίου όσο και του τελικού φαίνεται πως ε, είναι στο σωστό δρόμο. Τώρα για, τα, ε, για τις συμβάσεις του προσωπικού η κατάσταση είναι λιγότερο σοβαρή από ό,τι είχαμε προβλέψει και αυτό εν μέρη εξαιτία των υποστηρικτικών μέτρων που λάβαμε τόσο εμείς όσο και οι αρχές ε, της ε, Ολλανδίας. Αλλά ακριβώς και επειδή ε, αναλάβαμε δράση εγκαίρως. Ωστόσο, θα υπάρξει έντονη μείωση προσωπικού από το Μάρτιο του 2019. Γνωρίζουμε ότι θα χάσουμε περίπου 125 υπαλλήλου με συμβάσει ορισμένου χρόνου, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να μετακομίσουν μαζί με τον ε, οργανισμό. Ε, τώρα, η επικοινωνία το επικίνδυνο είναι η ζώνη της ε, κρίσης, δηλαδή από τη στιγμή ε, που πέσουν, ε, πέσει ο αριθμός του προσωπικού δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δουλειά μας και να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία ανθρώπων και ζώων. Ωστόσο, ελπίζουμε, και ελπίζουμε πώς θα καταφέρουμε να ε, ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό. Οι προσλήψεις ε, νέων ταλαντούχων ε, υπαλλήλων είναι μια επιλογή. Είχαμε περίπου 5.000 αιτήσει για θέσεις εργασίας και Συνεχίζεται αυτή η έντονη διαδικασία προσλήψεων. Βλέπετε ότι το γαλάζιο χρώμα ε, εδώ σημαίνει την πρόσληψη νέου προσωπικού. Το 2019 θα είναι μεταβατικό έτος, ε, κατά το οποίο θα ε, θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον και θα αλλάξει η εικόνα μας. Όπως βλέπετε θα χάσουμε πολλούς έμπειρους υπαλλήλου, αλλά καλωσορίζουμε και νέο ταλέντο με εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες ε, τις οποίες δεν είχαμε μέχρι τώρα. Θα είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ε, φέρνει μαζί του το μέλλον και αυτή η στρατηγική μας προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και στο σχέδιο που έχουμε υποβάλει στις δημοσιονομικές αρχές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων λοιπόν μπαίνει σε μία φάση ε, η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις τους ερχόμενους μήνες από τον Απρίλιο, αν όλα πάνε καλά, ή ε, το πολύ από τον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε ε, και θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Ωστόσο, το Brexit δεν είναι το μόνο που σκεφτόμαστε και δεν είναι το μόνο που μας απασχολεί αυτόν τον ε, καιρό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω για έναν αριθμό πρωτοβουλειών ε, πολύ ε, καλών που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τα φάρμακα για τα παιδιά, παιδιατρικά φάρμακα είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ κοντά σε όλους μας, η νομοθεσία ε, καθυστερούσε, ήταν στάσιμη για 10 χρόνια, αλλά έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη μελέτη των παιδιατρικών φαρμάκων. Τα φάρμακα πλέον έχουν ε, αλλάξει και από το 2007 έχουν εγκριθεί πάνω από 310 νέα φάρμακα ε, για, τα, για παιδιά, παιδιατρικά φάρμακα ε, το 1 τέταρτο όλων των νέων φαρμάκων που γκρίνονται είναι παιδιατρικά φάρμακα και η αλλαγές στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών για τα παιδιά, μολυσματικών, ρευματολογικών κτλ. είναι πολύ θετικές. Ο κανονισμός για, την, ε, τα παιδιατρικά φάρμακα έχει βελτιωθεί. Λαμβάνουμε και άλλα βήματα προς περαιτέρω βελτίωση. Για παράδειγμα, ε, βελτίωση του σχεδίου δράσης για, τα, για τον παιδιατρικό κανονισμό και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα σε δύο με τρία χρόνια. Επίσης, γνωρίζω ότι σας απασχολεί πολύ η ανθεκτικότητα και η μικροβιακή αντοχή. Ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας, γι' αυτό λοιπόν και καλωσορίζουμε το ψήφισμα το οποίο ενισχύει το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να στείλουμε, δηλαδή πως υπάρχει ανάγκη για επίγουσα δράση και πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ε, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίω, πρέπει να αναλάβουν δράση. Τα πράγματα δεν φαίνονται θετικά. Υπάρχει μία μείωση στην κατανάλωση αντιβιωτικών φαρμάκων από ε, ζώα κτηνιατρικών ε, αντιβιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η κατάσταση διαφέρει πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Η έκθεση SVAC που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα έχει περισσότερες λεπτομέρειες και βλέπουμε ότι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών κτηνιατρικών φαρμάκων είναι η αιτία για την μικροβιακή αντοχή, την αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις εξελίξεις αυτές, αλλά μπορούμε να την καθυστερήσουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε καθυστέρηση, ανάπτυξη νέων φαρμάκων και καινοτομία. Ε, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, όμως αυτό εξαρτάται από την χρήση των ε, φαρμάκων αυτών. Και εδώ έρχομαι στην καινοτομία. Χρειάζεται μια καινοτόμως προσέγγιση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Αυτή η καινοτόμως προσέγγιση δεν έχει ε, εμφανιστεί ακόμα, Όμω βλέπουμε κάποιες ενδείξεις πως ίσως αυτό αλλάξει στο μέλλον. Σίγουρα επίσης όλα αυτά χρειάζονται δέσμευση τόσο της βιομηχανία όσο και της πολιτικής. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο για να ε, κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεργαζόμαστε με ε, τους εταίρους μας, Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλους, έτσι ώστε να ε, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να ενθαρρύνουμε την βιομηχανία έτσι ώστε να αναπτύξει νέα ε, φάρμακα, να γίνουν κλινικές δοκιμές στα νέα αντιβιωτικά τα οποία θα είναι καλύτερα βελτιωμένα και θα αποφεύγονται διάφορες επιμολύνσεις όπως για παράδειγμα ρουλιμπόξ κτλ. Βέβαια, ο στόχος δεν είναι να μειώσουμε το βάρος της απόδειξης για τα νέα φάρμακα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης και αντιμετώπισης, το οποίο θα αντικαταστήσει τα τρία υπάρχοντα. Αυτό χρειάζεται βέβαια πολύ στενή συνεργασία με την ΕΦΣΑ και την ECDC, έτσι ώστε να εφαρμοστεί κατά γράμμα το σχέδιο δράσης το, για την ε, μικροβιακή αντοχή. Μετά, πρόσβαση στα φάρμακα. Είναι ένας μεγάλος τομέας ε, που απασχολεί ε, και εμάς και εσάς εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι να υπάρχει οικονομική ασφαλής πρόσβαση σε καινοτόμες ε, φαρμακευτικές αγωγές και θεραπείες. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε πολύ το ψήφισμα του 2017 ε, μας διαβεβαίωσε η Αρμόδια Επιτροπή, η Επιτροπή τότε πώς ε, θα μας βοηθήσει στο έργο μας, όμως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές προκλήσεις ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Ε, αμοιβή του ιατρικού προσωπικού, προκλήσεις σχετικά με τους ασθενείς, ε, πρόσβαση στην ε, θεραπεία. σε ό,τι αφορά τις αντικαρκυνικές θεραπείες με λεμφοκύτταρα κάρτη, υπάρχει τεράστια δυναμική να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην αντιμετώπιση των ε, διαφόρων ειδών καρκίνου. Όμως, αυτό βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι τομείς. Μετά, ε, τεχνολογία σύγκλησης. Εδώ χρειάζεται να εγκριθούν φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα που τα συνοδεύουν, το ε, λογισμικό που θα τα συνοδεύει, αλλά και ο τρόπος παράδοσης των ε, σκευασμάτων αυτών. Τα δεδομένα από όλα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται και να ταξινομούνται ίσως με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, προσβασιμότητας στα φάρμακα, της διαθεσιμότητας φαρμάκων τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει να δούμε τι ε, φάρμακα θα χρειαστούμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ε, παρασκευαστές κατανοούν το ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε τα δεδομένα που θα μας ε, μεταδώσουν να είναι αξιόπιστα ώστε να μας βοηθήσουν και εμάς το έργο μας, τη διαδικασία δηλαδή λήψης αποφάσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη νέων ε, κατηγοριών φαρμάκων. Γι' αυτό χρειάζεται μια ε, νέα μοναδική προσέγγιση η οποία θα μας πάει σε χαρτογράφητες ε, περιοχές στον χώρο της επιστήμης και της καινοτομίας. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία σε αρχικό στάδιο, έγκαιρη, και η βιομηχανία πρέπει να έχει επικοινωνία μαζί μας έτσι ώστε να ε, συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε επί του σχεδίου ε, δράσης και ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι το 67% των κλινικών δοκιμών δεν είναι κατάλληλες για χρήση όταν φτάνουν στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε επιστημονικά διότι δεν ε, επιτυγχάνουν τον στόχο και το 33% που ε, απομένει δεν αποτελεί καμία εγγύηση για να λάβει ένα φάρμακο έγκριση ε, προς διάθεση στην αγορά. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν αλλαγές, βελτιώσεις. Χρειάζονται επιστημονικά ε, δεδομένα τα οποία θα μας δείχνουν εάν ένα φάρμακο είναι ασφαλές αλλά και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει, δυνατό, υπάρχει περίπτωση αποτυχία, όχι γιατί ένα φάρμακο δεν είναι ενδεχομένω κατάλληλο, αλλά γιατί οι κλινικέ δοκιμέ δεν έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο. Στο 76% των κλινικών δοκιμών έχουν ένα κατάλληλο σχεδιασμό, είναι επαρκής ο σχεδιασμός, όμως έχουν ε, πιθανότητες αποτυχίες εξαιτία άλλων παραγόντων. Επίσης, ε, Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία κατάρτισης κλινικών δοκιμών ε, μέσω διαφόρων ε, φορέων τεχνολογικής αξιολόγησης ε, των σκευασμάτων όμως υπάρχουν διάφορα εμπόδια τα οποία φιλούνται στο φυστάμενο νομικό πλαίσιο. Συμπερασματικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χρειάζομαστε τις κατάλληλε δεξιότητε, την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πρέπει να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις ή έστω να τις ακολουθούμε κατά πόδας. Η μεταφορά του οργανισμού στο Άμστερνταμ θα συνοδευτεί από πολλές προκλήσεις και χρειάζεται λοιπόν να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο αυτή την αλλαγή αλλά και τις αλλαγές στην νομοθεσία. Ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξή σας ε, και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ταχύτητες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και όλων των πλασμάτων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας ε, στήριξε, να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μπιλιάννα Μπόρτσι, την Γενική Διευθύντρια, τον ε, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ματίας Γκρότε, τον κύριο Λαβία και εσάς κυρία Βαλεάν για την βοήθεια που μας έχετε δώσει, αλλά και τους κυρίους Μπιόρκ ε, και Λέμε, οι οποίοι εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράτη για την παρουσίασή σας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο σύνδεσμός Μάσα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων της Επιτροπής. Η κυρία Μπόζερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ράση, καλώς ορίσατε. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων εδώ και να πω ότι πραγματικά ελπίζουμε η μεταγκατάσταση του οργανισμού να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο της δημόσιας υγείας και έτσι ώστε να μην παρέμβουν, να μην παρεμποδίσουν την αποστολή του γεγονότα όπως το Brexit. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας μιλήσετε για ορισμένες ε, δραστηριότητες που θα προκύψουν μετά τη μετεγκατάσταση. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Θα επιθυμούσα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσον έχει ε, δοθεί μικρότερη προτεραιότητα σε ορισμένε ε, δραστηριότητες. Οι συνάδελφοι Κονέσκαρ, Μπάντεβαρ και Πεντιτζίνη έστειλαν μια γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα σχετικά με το θέμα της ικανότητα ε, του οργανισμού να λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια της φάσης μετεγκατάστασης. Εκφράσαμε κάποιο προβληματισμό ότι δεν έχει επαρκείς πόρους σε επίπεδο προσωπικού ο οργανισμός προκειμένου να μπορέσει να προετοιμαστεί για το Brexit και μας προβλημάτισε η ικανότητα της, ε, του οργανισμού να αντιμετωπίζει τρέχουσα νομοθεσία. Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίσουμε τι μέτρα παίρνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον οργανισμό να λειτουργήσει μετά την μετεγκατάστασή του. Μεταξύ των άλλων, ο Επίτροπος απάντησε ότι στα Έχοντας κατά νου τι του προπολογισμού του 19, το Ευρωπαϊκός Οργανισμός ζήτησε επιπλέον συμβόλαια και ε, αυτές οι πληροφορίες θα αναλυθούν από τις επιτροπές της Επιτροπής και ε, θα Θεωρήθηκαν όμως ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες για να μια αύξηση του προσωπικού ακόμα και ένα προσωρινό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο, μεγάλο του οργανισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε αίτημα αφορά την αύξηση του προσωπικού θα πρέπει να τεκμηριώνεται ορθά. Βεβαίω καταλαβαίνουμε τι προκλήσει με τι οποίε βρίσκεται αντιμέτωπο ο οργανισμό εν ώψη τη μετεγκατάσταση και καταλαβαίνουμε την πίεση που δημιουργεί αυτό για το ανθρώπινο δυναμικό. Πραγματικά μας εκπλήσει το ότι ο οργανισμός δεν υπέβαλε αιτήματα για ε, αιτιολογημένα για επιπλέον προσωπικό. Θα θέλαμε να μας δώσετε μερικές ε, εκ των έδω ό,τι αφορά την κατάσταση. Ο Ευρωπαίος Δήμο Μεσολαβητής πρόσφατα ξεκίνησε μία έρευνα ε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη φαρμάκων πριν ε, υποβληθούν τα ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό προκειμένου να δοθούν οι εγκρίσει. Ε, αυτές είναι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν επιστημονικές και ρυθμιστικές, ρυθμιστική παροχή ε, συμβουλών. Κύριε Ράζη, αναφερθήκατε στο ότι η επιστημονική γνώση βοηθάει αυτούς που παράγουν τα φάρμακα να υποβάλουν επιστημονικά δεδομένα και να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα προγράμματά τους δεν θα αποτύχουν γιατί δεν κατανοούν πλήρως ε, τις μελέτες ε, ή τις, ε, τους κανονισμούς. Είπατε ότι η επιστημονική παροχή συμβουλών δεν αποτελεί εγγύηση για μια θετική, για μια έγκριση κυκλοφορία στην αγορά. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, ε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες του διαμεσολαβητή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Λέμεν, ο οποίος είναι ανάμεσά μας σήμερα, να τον ευχαριστήσω που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τα τελευταία 12 χρόνια χρόνια. Συμμετέχει δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σα που ήρθατε σήμερα και να ευχηθώ και σε εσά και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ό,τι καλύτερο τους επόμενου μήνε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπόζεν. Τα μέλη έχουν τώρα το λόγο. Ήδη δύο εκδήλωσαν την πρόθεση να μιλήσουν. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά που βρίσκεστε ανάμεσά μας. Κύριε Διευθυντά, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο δυσάρεστο συμβάν της μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Φαρμάκων στο Άμστερνταμ και όχι στο Μιλάνο μετά το Brexit. Τώρα που έχει περάσει αρκετός χρόνος και κατά συνέπεια έχουμε μεγαλύτερη συνείδηση και μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι πολύ πιο σαφές αυτό που στην αρχή θεωρήσαμε μία λαϊκίστικη διαμαρτυρία, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχαν πραγματικ... ένας πραγματικός τεκμηριωμένος προβληματισμός για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Πεςτε μου λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το προαπαιτούμενο στην απόφαση της έδρας ήταν η παραγωγικότητα. Είναι αλήθεια ότι επιλέγοντας το Άμστερνταμ αποφασίσατε εν μέρη να ξεχάσετε το θέμα της λειτουργικότητας ό,τι αφορά θέματα αξιολόγησης ε, των αντικακινικών φαρμάκων, τα εισαγώγη φάρμακα, φάρμακα που δίνονται κατά την κοίηση. Και είναι αλήθεια ότι οι Ολλανδικές ε, αρχές ε, δεν υπευλήθησαν σε τριμερείς ελέγχους και αυτό είχε μία άμεση επίπτωση και σε άλλους ε, τομείς. Ξέρουμε ότι δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Είναι αλήθεια ότι το προσωπικό θα είναι επαρκές ε, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τις σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού βαρμάκων. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή, η οποία παρήσατε εδώ, αν αυτό είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, γιατί επιτρέψατε στους Ολλανδούς να πάρουν μέρος παρόλο που υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι. Γιατί επιτρέψατε ε, να γίνει αυτό ακόμα και όταν άλλαξε η προσφορά των Ολλανδών. Η δική μου ερώτηση είναι ποιοι είναι αυτοί οι Ολλανδοί. Μία χώρα που αρνείται να, ελε... να αλλά θέλει να, ε, ε, να, αλλά θέλει να ελέγχει. Μία χώρα που διακυβεύει ε, την ε, υγεία των Ευρωπαίων πολιτικών. Ένας προλογικός παράδεισος ζητάει μια διαδικασία κατεπίκουσα κατά της Ιταλίας. Στην ουσία δεν το ζητάει αυτό η Ολλανδία. Η Ιταλία θα ζητήσει ε, να εξεταστεί το θέμα νομικά. Η Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι από τις κατοχώρες. Και στο Άμστερνταμ φυσικά χαιρόμαστε πολύ που θα έρθει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμακών στην ε, χώρα μας. Γιατί όμως συνέβη αυτό, ε, διότι έχουμε πανεπιστήμια, Έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα και θέλουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία έτσι ώστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να γίνει λειτουργικό το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν πολλές ε, δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτήν τη μετακόμιση. Έχουμε έγκριτους επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι έχουν ε, κάνει αίτηση πρόσληψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Για μας ο συνάδελφος ο κύριος ε, Λαβή να πω ότι ήρθε, είδε με τα μάτια του ε, αυτό που κάνουμε και μπορεί να σας ε, επιβεβαιώσει όλα αυτά που σας λέω. Στο επίκεντρο για μας είναι η υγεία των Ευρωπαίων. Τώρα σε ό,τι αφορά την, την μικροβιακή αντοχή. Υπάρχουν πολλά ε, αποτελεσματικά φάρμακα, τα οποία όμως ε, έχουν υψηλό κόστος. Ε, εδώ πρώτο και κύριο μέλημα είναι το κέρδος των μετόχων. Ξέρετε, το θέμα όμως δεν πρέπει να είναι το κέρδος, αλλά να προσπαθήσουμε από κοινού ε, έτσι ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν τα κατάλληλα φάρμακα για τις ε, διάφορες παθήσεις. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα εγκρίθηκε και ένα ψήφισμα το οποίο ε, αφορά την αντιμετώπιση της βορελίωσης, της, του, της νόσου του Lyme. Και βλέπουμε ότι για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί χρειάζεται και ε, πολιτική βούληση, αλλά χρειάζεται και οι μέτοχοι να ε, παρατηθούν από ένα μερίδιο των κερδών τους. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με τη δική σας προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Ωραία. Εφόσον δεν επιθυμεί κάποιος το λόγο θα ε, ρωτήσω την Επιτροπή αν επιθυμεί να τοποθετηθεί. Όχι. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Μπιόρν Λέμερ, εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με ε, την κυρία Πόστανα και τον κύριο Ράση. Κύριε Λέμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό πιστεύω πως ε, ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Ράζη δηλαδή ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα μεταφερθεί στο Άμστερνταμ του χρόνου. Και δίχως αμφιβολία, ο κύριος Ράζη και το επιτελείο του έχουν καταβάλει τιτάνες προσπάθειες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις ε, δυσκολίες της μεταφοράς του οργανισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο στις κάτω χώρες. Προσπαθώντας ταυτόχρονα ε, να συνεχίσουν το έργο του οργανισμού για την ε, αντιμετώπιση νόσων. Αυτό που ανέφερε επίσης ο κύριος Ράζη είναι η μείωση του προσωπικού κατά περίπου 20%. Ε, αυτοί πάλι δεν θα μεταβούν στο Άμστερνταμ. Είμαι πεπισμένο όμως ότι ο κύριος Ράζη και το επιτελείο του θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω την εξή δήλωση ως πολιτικό όν και ως επιστήμονας. Κατά τη γνώμη μου το Brexit ήταν η πιο περιττή απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος της μεταφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων δεν ε, είναι μόνο τεράστιο, αλλά η πολιτική απόφαση για τη μεταφορά αυτή είναι μια καταστροφή, πολιτική καταστροφή, η οποία θα γίνει αισθητή για πολλά χρόνια. Ο οργανισμός ε, θα χάσει υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και αυτή η απουσία θα γίνει αισθητή τόσο σε εμά όσο και σε εσά. Και αυτό που θα χάσουμε επίση ε, είναι η συνεργασία ανάμεσα στου Βρετανού και του Ευρωπαίου συναδέλφου ε, σε διάφορα θέματα επιδημιολογία, ε, ιατρικών μελετών και άλλων. Τέλος, αυτή η έλλειψη συνεργασίας να γνωρίζετε πώς χτυπά τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ε, στο κέντρο του. Θα έχει επιπτώσει σε όλους. Είμαι πεπισμένος βέβαια ότι ο κύριος Ράζη και το επιτελείο του θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα αυτό, αλλά το θέμα αυτό ε, δεν είναι μόνο περιορισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit θα πλήξει και την επιστήμη. Σας ευχαριστώ. Πολύ εύστοχα τα είπατε, πολύ γλαφυρά. Θα πλήξει και την επιστήμη το Brexit και πολύ περιττή απόφαση. Έχουμε ε, επισημάνει και σε ψηφίσματά μας ότι το Brexit θα δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες παντού. Κύριε Ράση, παρακαλώ έχετε το λόγο για να απαντήσετε στα σχόλια και στις απορίες των συναδέλφων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από τις ερωτήσεις της κυρίας Μπίλιανα Μπόρζαν. Καταρχήν ρωτήσατε ποιες προτεραιότητες ε, θα δώσουμε και την προσέγγιση υιοθετούμε. Όπως ε, έδειξε και στη διαφάνεια, στην κόκκινη ζώνη βάζουμε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα και με τη διαδικασία έγκρισης και τη φαρμακοεπαγρύπνηση και, ε, και τον εντοπισμό των ε, δείξεων, δηλαδή αφορούν την ασφάλεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της, της διαδικασίας έγκρισης. Ε. Σε ό,τι αφορά τους σπόρους, ακριβώς επειδή θα έχουμε πρόβλημα πόρων, θα σταματήσουμε όλες τις νομοθετικές διαδικασίες. Ε, έχουμε ιατρική διαδικασία, τον γενικό κανονισμό ε, προστασίας δεδομένων και τον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Και δεν έχουμε για το GDPR και ε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν θα έχουμε εμπειρογνώμονες μόνο για το πρώτο θέμα θα έχουμε εμπειρογνώμονες, οπότε ξεπερνά τις ικανότητές μας. Γι' αυτό επισημάναμε το πρόβλημα. Ε, αυτό θα καθυστερήσει τις ε, νομοθετικές διαδικασίες. Μάλλον χάσαμε την ικανότητά μας να επιχειρηματολογούμε εύστοχα για την ανάγκη απόκτησης νέας εμπειρογνωμοσύνης. Τώρα το έχουμε διευκρινίσει, έχουμε ε, συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να έχει αποσαφινιστεί πια από πού προκύπτει αυτή η επιτακτική ανάγκη, η απεγνωσμένη ανάγκη αύξηση του προσωπικού μας. Δεν χρειαζόμαστε απλώ ε, τυχαίου υπαλλήλου, αλλά ειδικού εμπειρογνώμονε που να πληρούν ε, τις προποθέσει και να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουμε να ε, παρακολουθήσουμε αυτές τις νομοθετικές διαδικασίες. Τώρα, ξέρω ότι έχω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, και συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω και η Επιτροπή να πει στο Συμβούλιο για το πλέον προσωπικό μας ότι δεν, ε, δεν μετράμε κεφάλια ε, και δεν χρησιμοποιούμε συμβασιούχους όταν πρέπει να χάσουμε το μόνιμο προσωπικό. Απλώς υπάρχει μια τριετή μεταβατική περίοδο για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες. Οπότε, σε τελική ανάλυση δεν θα αυξήσουμε το προσωπικό μας, αλλά θα το μειώσουμε. Και μάλιστα, ε, προσωρινά μειώνουμε την απώλεια του προσωπικού. Και αυτή τη στρατηγική θέλω να σας παρουσιάσω και στην αρχική μου ομιλία. Στο μέλλον, αυτό που θα παρουσιαστεί ίσως δεν ε, καλυφθεί από τους ε, ε, εμπειρογνώμονες που έχουμε. Οπότε, με τη μετακόμιση θα έχουμε πρόβλημα όχι μόνο με τη μείωση προσωπικού, αλλά θα έχουμε και με την ευκαιρία να προσλάβουμε τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες για την επόμενη πενταετία ή δεκαετία, για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Αν συμφωνήσετε με την έγκριση αυτών των επιπλέον 40 υπαλλήλων, φορέων γνώσης όπως λέμε, ε, όσους δεν θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε άμεσα ή θέλουμε να προσλάβουμε άμεσα, θέλουμε να ανταποκριθούμε στο νέο κύμα το ορμοθετικό που έρχεται. Και παραλαμβάνω, οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξέλιξεις ε, συντελούνται με ταχύτητα του φωτός. Θέλουμε λοιπόν ε, όχι απλώς να αντικαθιστούμε τους χαμένους υπαλλήλους ένα προς έναν, αλλά να τους αντικαθιστούμε με κατερτισμένους, μορφωμένους και με τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη επιστήμονες. Και γι' αυτό θέλουμε την υποστήριξή σας για να γίνει δεκτό το αίτημα για την στελέχωση με 40 ε, νέα μέλη του ΕΟΦ. Σε ό,τι αφορά τη διαμεσολαβήτρια. Ναι, καλωσορίζουμε τις ε, νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της Έμιλι Ράιλι, για να διευκρινίσουμε περαιτέρω την κατάσταση και ήδη στην παρουσίασή μου σας έδωσα κάποια βασικά στοιχεία και θα ήθελα να διασκεδάσω κάποιες εμβολίες ή να ξεκαθαρίσω κάποιες παρεξηγήσεις. Δεν κάνουμε ανάλυση δεδομένων μαζί τους. Εμείς εξετάζουμε τα δεδομένα και λέμε στους επικριτές, όχι στη διαμεσολαβήτρια, στους ε, επικριτές, λέμε ότι δώστε μας την ευκαιρία για να διαλύσουμε αυτές τις παρανοήσεις που δημιουργήθηκαν. Εμείς ε, αναλύουμε το σχέδιο ανάπτυξης, καθορίζουμε ποιο είναι το καλύτερο σχέδιο ανάπτυξης για να υλοποιήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ήδη μελέτη και δεδομένου ότι η μελέτη για την στατιστική ισχύ και τις κλινικές ε, αποδείξεις που χρειάζονται ε, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Αν φτάσει σε αυτό το μαγικό στάδιο, ίσως λάβει την έγκριση και κάποιοι άλλοι ε, χρόνια ολόκληρα μετά θα αξιολογήσουν τα στοιχεία. Οπότε δεν υπάρχει σύγκρουση φερόντων, δεν υπάρχει συνέχεια και εμεί θέλουμε να εξασφαλιστεί κάποια συνέχεια και κάποια συνέπεια και συνοχή της διαδικασίας. Πάντως η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ διαφορετική από την συμβουλευτική διαδικασία, που επίσης είναι θελοντική δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για την λήψη τέτοια επιστημονικής γνωμάτευσης. Είναι μια ευκαιρία. Αυτό που, προέχει είναι να γίνονται σωστέ κλινικές δοκιμές χάρη του ασθενού. Γιατί αυτό είναι ο κίνδυνο και η ντροπή μια κλινική δοκιμή που γίνεται να μην οδηγήσει πουθενά να μην τελεσφορήσει. Φυσικά, αν πώς θα έχουμε πιο αποτελεσματική διαδικασία. Καλύτερες μελέτες, καλύτερα αποτελέσματα και επιτυχημένες κλινικές δοκιμές. Και αυτό θα είναι επιτυχία και για τον ασθενή και για τον ε, ρυθμιστικό φορέα και για τον επενδυτή ότι έκανε σωστές επιλογές. Και να προσθέσω και ένα στοιχείο που δεν παρέλειψα προηγουμένως. 30% των ε, ε, σχεδίων που έρχονται στο σχέδιο Prime για τα κατά προτεραιότητα φάρμακα ε, αποφασίζουν σε κάποια φάση να σταματήσουν το σχέδιο ανάπτυξης γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν πάει πουθενά. Και λαμβάνουν υπόψη και τη δική μας ανησυχία για τον ασθενή πριν περάσουν στην κλινική δοκιμή. Έτσι θέλουμε καλύτερα στοιχεία και φροντίζουμε γι' αυτό και ασφαλέστερα στοιχεία σε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρόκειται να τη χάσουμε και θα το πούμε στην έρευνα που διενεργεί η διαμεσολαβήτρια, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ε, ο Δ. Πεντιτσίνη με έθεσε κάποιες ερωτήσεις, μερικές όμως ε, ε, είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Για τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η διαδικασία κατάρτισης των προτεραιοτήτων μας πιστεύω ότι είναι χρηστή, στιβαρή και διέπεται από τη μέρημνα για τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι ο γνώμονάς μας, η δημόσια υγεία και η κόκκινη γραμμή μας. Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία και συνεχώς ασκούμε πιέσει στις Ολλανδικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και η δική μας ιεραρχία προτεραιοτήτων αφορά περισσότερο την απώλεια προσωπικού και όχι το θέμα της επιχειρησιακής συνέχειας λόγω της ε, μετεγκατάστασης του οργανισμού. Θεσμικά, δεν πρόκειται να κάνω σχόλια, και εγώ Ιταλός είμαι και έχω διπλό λόγο να μην επεκταθώ, να σιωπήσω στο σημείο αυτό. Πάντως θεσμικά πιστεύω η προτεραιότητα οφείλεται, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων οφείλεται στην απώλεια προσωπικού λόγου της μετεγκατάστασης. Και στην κυρία Σρέερ Πίρικ, κάπως έτσι. Δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας σίγουρα. Πάντως, ε, αισθενιζόμαστε τον προβληματισμό σας για την τιμολόγηση ε, οι τιμές των φαρμάκων είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και τις σημαντικότερες ανησυχίες μας τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορούμε να εγκρίνουμε φάρμακα σε προσιτές τιμές. Βέβαια δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, παρόλο που υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε το όσο πιο αποτελεσματικό περιβάλλον γίνεται για να διευκολύνουμε τους αρμόδιους ε, για τις διαπραγματεύσεις να προτείνουν ευνοϊκότερες τιμές αυτές τις διαπραγματεύσεις ώστε η ανάπτυξη φαρμάκων να γίνεται σε ένα πιο αποτελεσματικό περιβάλλον και άλλο το φάρμακο να διατίθεται σε πιο προσιτές τιμές. Επίσης προσπαθούμε με τις δοκιμές να δώσουμε τις ε, τα καλύτερα στοιχεία στα σώματα ε, αξιολόγησης των ε, τεχνολογιών υγείας για να μπορούν να εντοπίζουν την προστιθέμενη αξία της κάθε καινοτόμους πρότασης. Πάντως θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η κλινική προστιθέμενη αξία και ποια η καθολική προστιθέμενη αξία. Γιατί όταν προσφέρουμε κάποια θεραπευτική προσέγγιση, ε, μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η κλινική προσθέμενη αξία είναι καθολική, είναι οικουμενική αξία. Οπότε κάνουμε αξιολόγηση και αυτών των στοιχείων και συνεργαζόμαστε με τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, τους HTA, και θέλουμε να εξορθολογήσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία χάρη στην ευπρόσδεκτη πρόταση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Αυτά μόνο μπορούμε να κάνουμε ως προς τις τιμές των φαρμάκων. Και για την επιστημονική γνωμάτευση, αν ο φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας ε, μας πλησιάσει, μπορούμε να το πούμε τι μπορεί να ρωτήσει και τι να μην. Και αυτό ε, σε ό,τι αφορά το συγκριτικό σκέλος ε, συνιστά μεγάλη πρόοδο και για τον ε, ασθενή και για τον φορολογούμενο και για τις φαρμακοβιομηχανίες που ξέρουν από την αρχή τι πρέπει να παρασκευάσουν και δεν έχουν καμία ε, δικαιολογία, γιατί ξέρουν τι αποδείξα θα πρέπει να δώσουν και μάλιστα εγκαίρως. Ό,τι αφορά την έρευνα για τη βορελίωση, την όσο του Λάιμ, φυσικά και εκτιμώ ιδιαίτερο την ε, ανάγκη Δημόσια έρευνα, έρευνας με δημόσια κονδύλια, όταν δεν υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον για τη διενέργεια τέτοια ε, έρευνα. Βέβαια, εμεί δεν είμαστε ερευνητικό κέντρο και χαίρομαι που στο νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προβλέπονται αρκετά κονδύλια για την έρευνα και στον τομέα των λιμωδών ε, νόσων και ίσως ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, Φαρ... Φαρμάκων θα έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει. Και η δυνατότητα να έχουμε οικονομικούς πόρους, ε, τώρα που έχουν αρθεί τα εμπόδια, ε, θα προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε την έρευνα προς τις ε, ιατρικές ανάγκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Λέμερ για τα ευγενικά του λόγια. ελπίζω να τα καταφέρουμε, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, πάντως προσπαθούμε και κάνουμε το πάντα δυνατόν. Και ευχαριστώ για τη στήριξη και τις καλές σας συμβουλές όλα αυτά τα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση και μετά θα περάσω στο τελευταίο σημείο τη ημερησία διάταξη. Καταρχά θα έχουμε ένα εργαστήριο για τον εγκέφαλο και νέα προσέγγιση στις εγκεφαλικές νόσους. Το, το έχει οργανώσει η Επιτροπή μας. Ο κύριος Πέτρελ και η κυρία Καπεζόν είναι οι συμπρόεδροι. Αυτό το εργαστήριο θα γίνει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου από τις 10 και μετά και θα σας έλεγα να πάρετε μέρος. Σε όση διαφορά αφορά τον τελευταίο τριμερή διάλογο που αφορά την Επιτροπή μας, θα αναφερθώ και σε αυτό το θέμα. Ο δεύτερος άτυπος τριμερής διάλογος για τα αυτοκίνητα και το διοξίδιο του άνθρακος έγινε συζήτηση τώρα σε ό,τι αφορά λιγότερα πολιτικά θέματα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των έξι ετών. Ε, τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα επετεύθη ο ε, συμβιβασμός σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Επιπλέον ημέρα θα πρέπει να συζητηθούν στον επόμενο τριμερή διάλογο. Σε ό,τι αφορά περισσότερο πολιτικά θέματα, ε, μηδέν εκπομπές ε, του άνθρακα, εξαιρέσεις, ανάλυση κύκλου ζωή, ανάλυση κύκλου ζωής, καινοτομίε. Οι δύο συνομοθέτε θα πρέπει να υποβάλουν τροπολογίες εάν θέλουμε επιτευχθεί ο συμβιβασμό και να επιτευχθεί πρόοδος στην τρίτη συνάντηση που προβλέπεται και τις 4 Δεκεμβρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, εκθέση για το περιβάλλον, έγινε η πρώτη τριμερή συνάντηση Είχαμε μία, υπήρξε μία ανταλλαγή απόψεων. Παρουσιάσαμε την άποψή μας για την πρόταση της Επιτροπής. Οι συζητήσεις έδειξαν ότι οι συνομοθέτες ακολούθησαν μία παρεμφερή προσέγγιση για μία σειρά από θέματα με εξαίρεση κυρίως το άρθρο T και τις διατάξεις που αφορούν την Επιτροπολογία. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να αφήσουν τα θέματα αυτά για εξέταση σε τεχνικό επίπεδο με στόχο να επαναξεταστούν στην επόμενη τριμερή συνάντηση που θα οργανωθεί στο μέλλον. Δεν έχουμε ακόμα ε, ημερομηνία στο εγγύς μέλλον. Τώρα, το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης για σήμερα αφορά μια πρόταση ψηφίσματος για μία αντίρρηση για την έγκριση ορισμένων χρήσεων του διχρωμικού νατρίου. Εντάξει, σωστά το, πρώτη, το πρόφερα. Ο κύριος Μπέιγα, αλλά υπάρχουν και μερισμένοι συνεισηγητές. Νομίζω ότι όλους θα τους εκπροσωπήσει ο κύριος Αικάουτ. Ε, Κύριε Αικάουτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου που πήραν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ελπίζω να μην καταδεικνύει αυτό τη σημασία του, τη βαρύτητα του θέματος, γιατί πρόκειται για μια χημική ουσία που ενδεχομένως γνωρίζουμε από την ταινία «Έρινε Μπρόκοβιτσα. Είναι γνωστό λοιπόν αυτό το σχέδασμα. Είναι περίεργο το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα Έχω να κάνω μερικέ σημαντικέ ερωτήσει στην Επιτροπή. Αν κοιτάξω τι πληροφορίε που υπάρχουν και αν διαβάσετε τι ε, γνωμοδοτήσει που αφορούν την αξιολόγηση κινδύνων, φαίνεται ότι το θέμα είναι απόλυτα σαφέ, απόλυτα ξεκάθαρο. Δυστυχώ ε, δεν βλέπουμε τις προτάσεις από την Επιτροπή και γι' αυτό το λόγο είχαν ε, αντιρρήσεις και υπάρχει μια αντίρρηση στην απόφαση αυτή. Αν διαβάσετε την αξιολόγηση ε, ΡΟΚ της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου αναφέρεται σαφώς ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτότητα καθορισμού του επίπεδου της ουσίας. Είναι ιδιαίτερα καρκινογόνος και θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις οποιαδήποτε έκθεση. Εάν διαβάσετε το ρίτσα διαπιστώσετε ότι είναι απόλυτα σαφές. Το ρίτσα αναφέρει ότι αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα και εάν δεν έχει επιπτώσεις θα πρέπει να δει κανείς αν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και κατά πόσων προκύπτουν κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δοθεί άδεια. Το ρίτς είναι πάρα πολύ σαφές εδώ. Δυστυχώς, η Επιτροπή προτείνει ε, μια έγκριση και το επιχείρημα είναι ότι στην αρχική διαδικασία δεν υπήρχαν γνωστές εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή θα κρυφτούν πίσω από διαδικαστικά επιχειρήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι ο ΙΕΚΑ αξιολογεί τους κινδύνους και η Επιτροπή διαχειρίζεται τους κινδύνους ακόμα και αν η ΕΚΑ που γνωρίζουμε ότι εξέτασε το θέμα αυτό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ορισμένα θέματα που αφορούσαν την ποιότητα του αιτήματο. Παρόλα αυτά όμως το αξιολόγησαν, ζήτησαν διαβουλεύσεις ε, για το αν η υπάρχουν εναλλακτικέ. Ε, είπαν λοιπόν ότι κανένα δεν απάντησε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ και συνεπώ δεν υπάρχουν. Ήταν γνωστό στην Επιτροπή ότι υπήρχαν εναλλακτικέ λύσει. Ε, η Επιτροπή λοιπόν ε, λέει ότι διαβάζουμε ότι μας δίνει η ΕΚΑ και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Τότε αν συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε την Επιτροπή. Τότε βάζετε τη βούλαν σε αυτό που λέει η ΕΚΑ και τελειώσαμε. Όχι. Η Επιτροπή λέει ότι εκείνοι είναι οι αξιολογητέ, εμεί είμαστε οι διαχειριστέ του κινδύνου. Νομίζω ότι τα θέματα είναι πολύ απλά τώρα για την Επιτροπή. Συμφωνείτε ότι το διχρωμικό νάτριο είναι μια ουσία την οποία δεν υπάρχει κατόφλια. Συμφωνείτε ότι το ρίτσι είναι απόλυτα σαφές ότι δεν θα πρέπει να δοθεί έγκριση εάν υπάρχουν εναλλακτικέ ουσίε. Συμφωνείτε ότι οι τελευταίες πληροφορίες καταδεικνύουν ότι υπάρχουν εναλλακτικέ ε, ουσίες. Τότε το ερώτημα είναι γιατί συνεχίζετε να, να διοδοτείτε και αυτό ε, σε αντίθεση με τις βασικές αξίες του Ρίτσε. Πέρα, χωρίς τα επιχειρήματα ε, του τι κάνει η ΕΚΑ, γιατί εσείς ως Επιτροπή, τον πολιτικό ρόλο, να υποβάλλετε πρόταση και αυτό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στους κανόνες ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση. Και για το λόγο αυτό εμείς υποβάλαμε μία αντίρρηση σε αυτή την πρόταση και ελπίζουμε ότι η πλειοψηφία στην Επιτροπή αυτή θα συμφωνήσει προκειμένου να προκύψει μία σαφής δήλωση από το Κοινοβούλιο πριν να αποφασίσουν ε, οι χώρες μέλη. Είναι εφαρμοστική πράξη, συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζει το Κοινοβούλιο πριν να αποφασίσει το Συμβούλιο. Γι' αυτό θα θέλαμε να το τον υποβάλουμε στη μήνυ Ολομέλη την επόμενη εβδομάδα στο Νοέμβριο για να κάνει τη δουλειά το Κοινοβούλιο πριν ε, ε, περάσει το θέμα στο Συμβούλιο. Νομίζω όμως το, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην κρύβεστε πίσω από διαδικαστικά επιχειρήματα της ΕΚΑ γιατί εδώ μιλάμε για καρκινογόνους ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει ουδός, δεν υπάρχει κατόφλι και αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, οι κανόνες είναι απλοί δεν θα πρέπει να δοθεί άδεια. Ε, μίλησα λίγο περισσότερο, ε, ε, αλλά νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για να απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές. Έχω την, τα λόγια του κύριου Μπουσόη, σκιώδη εισηγητή από το ΕΛΚ, και επειδή η πτήση συναδέλφου καθυστέρησε θα διαβάσω εγώ τις παρατηρήσεις του. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την παρούσα ένσταση. Ο Ετών λοιπόν υπέβαλε αίτηση επανασυσκευασίας του διχρωμικού νατρίου για σκοπό βαφής ε, μαλλιού σε, για βιομηχανικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού. Παρά το γεγονός ότι τα άρθρα 55, 64 και 62 του κανονισμού REACH αναφέρουν ότι ο ετών θα πρέπει να παρέχει το μέσο της αντικατάσταση καθώς και εναλλακτικέ λύσεις έτσι ώστε η Επιτροπή RAC να αξιολογήσει αυτά τα στοιχεία. Από την άλλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σύστησε να δοθεί η έγκριση υπό προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον ληφθούν μέτρα διαχείρισης κινδύνου και επιπλέον ορισμένες ε, κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Έχουν συγκεκριμένη πολιτική που δεν επιτρέπουν τη χρήση του διχρωμικού νατρίου για την ε, υψηλή ραπτική. Χρησιμοποιούν χρωστικές ουσίες οι οποίες παράγονται με πιο ασφαλή τρόπο. Ε, τούτου λεχθέντος λοιπόν η θέση του σχεδίου του ΕΛΚ είναι να ούτε να στηρίξει ούτε να απορρίψει την ένσταση αυτή, αλλά να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διαδικασία της έγκρισης, έτσι ώστε να λάβει τη σωστή απόφαση χωρίς να ε, δυσχεράνει τη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως θα ήθελε να εκφράσει και ο ίδιος τις ε, ανησυχίες του. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη του κύριου Μπουσό για την ένσταση. Ε, κυρία Κάντενμπαχ, θα θέλετε το λόγο. Περνώ κατευθείαν στους κοιόδης ηγητές. Ε. Ναι, θα ήθελα και εγώ λοιπόν να πω τα εξή. Σε μια που ο Παύλ Πόκ είναι συνεισηγητή των σοσιαλδημοκρατών, θα μιλήσω εξ ονόματό του και εμεί στηρίζουμε απόλυτα τα όσα είπε ο Μπα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Γενική Διεύθυνση Γκρό, τον κύριο Κάρλο Πετινέλη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να τοποθετηθείτε στις ανησυχίες που εκφράζουν οι εισηγητής και οι συνεισηγητές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω πως δεν ονομάζομαι Πετινέλη, αλλά Fluent είμαι διευθυντής ε, για... και αρμόδιος των κανονισμών REACH στη Γενική Διεύθυνση GROW. Με συγχωρείτε, λέει πρόεδρο, αυτές τις πληροφορίες έχω λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ε, καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε. Ε, οι πληροφορίε που λάβατε είναι σωστές, όμως ε, θεωρούσαμε ότι το σημείο αυτό θα εξεταστεί λίγο αργότερα. Και ε, θα μιλήσω λοιπόν εξ ονόματος του διευθυντή μου, του κύριου Πετινέλη. Είμαι επικεφαλής για θέματα που αφορούν το κανονισμό Ρίτσο, όπως σας είπα. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας δώσω το πλαίσιο στο οποίο ε, κινείται αυτή η ένσταση. Η αναθεώρηση του κανονισμού Ρίτσο, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2018 και συζητήθηκε στην Επιτροπή σας, αναγνωρίζει ότι η διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με τον ε, κανονισμό REACH χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Η σημασία της έβρεσης εναλλακτικών λύσεων έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι περισσότερες επικίνδυνες ουσίες ή ουσίες, ιδιαίτερα ανησυχητικές ουσίες. Στηρίζουμε επίσης την ανάγκη καλύτερης χρήσης της πληροφορίας και της δημόσιας διαβούλευσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ο ΕΚΑ, οι διάφοροι από τα κράτη-μέλη και άλλοι αρμόδιοι φορεί συνεργάζονται έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δράσεις και να υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων μέτρων. Η πρόταση ψηφίσματος αναφέρεται στις ελλείψεις που έχουν προκύψει μετά από την ανάλυση μας για στην διαδικασία έγκρισης από τον συνάδελφο Ομερτσάνο αναφέρεται στην διαδικασία ΤΣΕΑΚ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την έλλειψη συγκέντρωσης κατάλληλων στοιχείων και ε, εναλλακτικών λύσεων κατά την διαδικασία έγκρισης από την εταιρεία Grupo Κόλια. Η αιτιολόγηση είναι ότι υπερβαίνει τις αρμοδιότητες που δίνει ο κανονισμός REACH. Τώρα, η ΣΕΑΚ έχει επιβεβαιώσει την τεχνική και οικονομική ε, δυνατότητα τόσο στην ε, περίπτωση που αναφέρα όσο και στην περίπτωση Ιλάριο Ομερτσάνο. Και οι δύο εταιρείες υπέστησαν εξέταση και ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και είδαμε και στις δύο περιπτώσεις ε, ότι η πρόταση δεν είναι εφικτή. Ε, προτείναμε αναθεώρηση σε 7 έτη. Κατά την κατάρτιση της, ε, του σχεδίου απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήσαμε και με τα κρατημέλη και με την Επιτροπή για τον κανονισμό REACH και το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκε η Επιτροπή μας είναι ότι δεν είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικών λύσεων από τις δύο αυτές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε βασίσει την απόφασή μας σε αυτό. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που εντοπίστηκε οδήγησε στους συναδέλφους μας το να μειώσουν την ε, περίοδο αναθεώρηση από τα 7 στα 4 έτη. Αυτή η πρόταση υπερψηφίστηκε από μια ειδική πλειοψηφία στην Επιτροπή «Ριτς», και πέρασε στην δική σας επιτροπή μετά. Και στις δύο περιπτώσεις, και στον Κρουποκόλλη και στον Λάριο Μερτσάνο, υπάρχουν πολλές ομοιότητες και θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να εθετήσουμε μια ενιαία προσέγγιση που θα επιτρέπει σε βραχή χρονικό διάστημα να διεξαχθούν όλες οι αξιολογήσεις. Γι' αυτό λοιπόν προτείναμε και μια πιο σύντομη περίοδο αναθεώρησης. Για τους λόγους αυτούς έχουμε προτείνει τόσο και στην περίπτωση Λάριο Μερτσάνο να εγκρίνουμε περίοδο αναθεώρησης μόνο 4 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δράσει πλήρως συμμορφούμενη με τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω, μια και έχουμε χρόνο, αν θέλετε να επανέλθετε κυρία Εκχαουτ. Όχι, από ό,τι φαίνεται, οπότε ολοκληρώνουμε η συζήτηση και μάλιστα θα ψηφίσουμε για αυτή την αντίρρηση αύριο το πρωί. Κατά πάσα πιθανότητα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αυτά για σήμερα το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση. Ραντεβού αύριο το πρωί με τις ψηφοφορίες. Καλό βράδυ.